Varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Vi har en eh, intressant... Καλώς ορίσατε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε μία ενδιαφέρουσα ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα, αλλά και για αύριο. Καλώς ορίζω θερμά όλους τους παρόντες και θα ήθελα να χαιρετήσω ιδιαίτερα και ορισμένους νέους Σουηδούς ε, που έχουν έρθει για να παρευρεθούν στις εργασίες της Επιτροπής μας. Επειδή είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά από τη γιορτή της γυναίκας, Δράτω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και την εξαιρετική μας γραμματεία για τη συνεργασία τους κατά τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας. Οι προβληματικές μας είχαν την πρωτοκαθεδρία τη μέρα εκείνη. Εμείς ε, ελπίζουμε να έχουμε ε, μεγάλη υποστήριξη και στο μέλλον ε, για, τις, για τους αγώνες μας. Ευχαριστώ λοιπόν που προωθήσατε διεθνώς ε, τα θέματα που αφορούν στις γυναίκες. Πάμε στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει μία μικρή αλλαγή στο σημείο 8. Συζήτηση με την κυρία Λάντμπακ, τη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, θα συζητηθεί στο 9. Δηλαδή η κυρία Φραντσέσκα Μπαλτζάνη, η συγγήτρια για τον προπολογισμό του 2012 θα πάει στο σημείο 8 και η κυρία Λάντμπακ πάει στο 9. Αυτό οφείλεται στα ωράρια ταξιδιού της κυρίας, της κυρίας Λάντμπακ. Αν δεν έχετε αντιρρήσει στην ημερήσια διάταξη, έτσι όπως την προτείναμε, εγκρίνεται ανακοινώσει της Προέδρου στο σημείο 2. Λοιπόν, 24 Μαρτίου από τις 9 μέχρι τις 10 και μισή θα έχουμε μία έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τον Μισελ Μπασλέ στις 24 Μαρτίου από τις 9 μέχρι τις 10.30. Με την κυρία Μπασλέ θα συζητήσουμε. πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 13ης Δεκεμβρίου 2010, 20 Ιανουαρίου 2011, 26 και 27 Ιανουαρίου του 2011. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο φάκελό σας. Θεωρούμε εγκεκριμένα τα πρακτικά γιατί δεν λάβαμε παρατηρήσεις. Πάμε στο σημείο 4. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τη Γιούτα Χάουκ που είναι πρόεδρος της ειδική Επιτροπής σχετικά με τις ε, προκλήσεις πολιτικής ε, και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη ένωση μετά το 2013. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που υποδεχόμαστε την κυρία Χάουκ για να μας ενημερώσει και εμείς με τη σειρά μας θα τις υποβάλουμε τις προτάσεις μας και τις ιδέες μας. Θυμίζω ότι οι συντονιστές της Επιτροπής μας αποφάσισαν να συνεισφέρουν σε αυτή την έκθεση παρουσιάζοντας ε, τροπολογίες ε, στην Ειδική Επιτροπή. Θα σας δώσω το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας στο τέλος της συζήτησης. Κυρία Χάουγκ, έχετε το λόγο. Ja, ähm, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην Επιτροπή σας. Είναι πολύ θετικό λοιπόν στο βαθμό του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας να μπορώ να εκφράζω ως ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ αυτά τα οποία έχουν λάβει η χώρα στη δική μας Επιτροπή. Ξέρετε ότι ξεκίνησαμε πέρσι μετά το, τις καλοκαιρινές διακοπές και έχουμε χωρίσει την εργασία μας σε τρία τμήματα. Η πρώτη φάση αφορούσε τις εργασίες μας. Αφορούσε τα γενικότερα πολλές φορές τεχνικά θέματα. Δηλαδή, καταρχήν, ποια θα έπρεπε να είναι η διάρκεια της επόμενης <clears throat> περίοδου δημοσιονομικής σχεδίασης. Η δεύτερη φάση, η οποία ξεκίνησε μετά τα Χριστούγεννα, το 2010 συγκεκριμένα, αφορούσε την απασχόληση με επιμέρους τομεακές πολιτικής, αγροτικά θέματα, θέματα συνοχής, θέματα εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία παίζουν κάποιο ρόλο στον προϋπολογισμό μας και την πρόσφατη βδομάδα στο Στρασβούργο, την Πέμπτη, κάναμε την τελευταία μας συνάντηση σε σχέση με το θέμα αυτό <clears throat> και στη συνέχεια μάλλον σε αυτή την τελευταία συνάντηση ασχοληθήκαμε με τα θέματα εσωτερικών και μετανάστευσης και στη συνέχεια το ερώτημα του πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, σημαντικότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού. Είμαστε λοιπόν ενώπιον σημαντικών προκλήσεων αλλά συγχρόνως υπάρχει μεγάλη σύμπνοια μεταξύ μας <clears throat> σε σχέση με τις ακολουθητές πολιτικές, όχι μόνο τώρα αλλά και στην επόμενη περίοδο δημοσιονομικών πρόπτικών. και η Στατηγική Ευρώπη 2020 έχει προταθεί από την Κομισιόν, έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρσι εκδώσαμε ένα ιδιαίτερα θετικό ψήφισμα για αυτή τη στρατηγική. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία ζητούμε για τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις και φυσικά πάντα το ερώτημα είναι ποιε θα είναι οι πολιτικέ οι οποίε προσφέρουν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και πω μπορούμε τα κονδύλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα με το πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να τα χρησιμοποιήσουμε και εξάλλου με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την σύνδεση μεταξύ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών. Πώς θα διαμορφώσουμε λοιπόν ένα ενιαίο σύνολο ενεργειών. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μας απασχόλησαν στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ και βλέπετε τώρα και στον φάκελό σας το έγγραφο της Επιτροπής μας που περιέχει το εισηγητικό μας σχέδιο. Προς το παρόν είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκε στις μεταφραστικές υπηρεσίες και πιστεύουμε ότι μεθαύριο το αργότερο θα είναι διαθέσιμο το σχέδιο αυτό σε όλες τις γλώσσες. Αυτά λοιπόν τα οποία προτείνει ο, εισαγγελ... ο εισηγητής μας, ο κύριος Γκαριγά. Όλα αυτά είναι το περιεχόμενο της έκθεσής μας και που πιστεύω ότι αντανακλούν ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα οποία συζητήσαμε στην Επιτροπή Σούρε. Και όταν αναφέρομαι στην Επιτροπή Σούρε δεν αναφέρομαι μονάχα στους ε, στα μέλη της Επιτροπής αυτής της έκτακτης Επιτροπής, αλλά και στους εκπροσώπους των ε, επιτροπών, των υπολείπων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τους προσκαλέσαμε όταν συζητεί κάποιο θέμα της αρμοδιότητας των επιτροπών τους. Αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε στην επόμενη περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σωστές προοπτικές και έναντι του Συμβουλίου αυτό φυσικά θα απαιτήσει μια μεγάλη πλειοψηφία, μια ευρεία πλειοψηφία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μην περιοριστούμε σε ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο, αλλά να μπορέσουμε να παίξουμε και ένα αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των προοπτικών. Θα συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή Σούρε το πώ ακριβώ θα προχωρήσουμε σε διαδικαστικό επίπεδο. Φυσικά θα συζητήσουμε την πρόταση του εισηγητή σε σχέση με την τελική έκθεση τη Επιτροπή μα, αλλά πρέπει περαιτέρω να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να κινηθούμε ώστε το Συμβούλιο τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του Συμβουλίου να πιστεί από τα επιχειρηματά μας για την πρέπουσα διαμόρφωση των, δημοσιονομικών προοπτικών για το επόμενο διάστημα και να ακολουθήσει τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Αυτό φυσικά δεν είναι τόσο απλό. Είδαμε ήδη από την διαδικασία του προϋπολογισμού του 2011 ότι υπήρξε μια στάση <clears throat> απόλυτης άρνησης από την πλευρά του Συμβουλίου να συζητήσει θέματα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα οποία έλκονται από τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Εμείς όμως έχουμε απόλυτη επίγνωση αυτά, αυτών τα οποία λέει η συνθήκη της Λισαβόνας και βλέπουμε ότι η συνθήκη αυτή δίδει ορισμένες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς θέλουμε αντίθετα από τη στάση εμπλοκής του Συμβουλίου να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αρμοδιότητες. Όπως ξέρετε, δόξα το Γιαραμπή, τα πράγματα δεν πήγαν τόσο άσχημα τελικά στο, στα θέματα του προπολογισμού το, τον περασμένο χρόνο και οι επερχόμενες προεδρίες συμφωνούν απόλυτα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζήτηση για τις ε, επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους και όλες μας ότι το Συμβούλιο θα πρέπει μεν ομόφωνα να αποφασίσει για αυτήν την, αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά με την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το κομβικό σημείο, αυτό είναι το σημείο στο οποίο είπαμε εμείς ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα πάλι όπως είχαν γίνει τα προηγούμενα δέκα χρόνια, να καταλήγουμε σε νύχτες των μακρών μαχερών, όπως ελέγεται. <clears throat> Δεν έχει νόημα να τσακωνόμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα και μόνο την τελευταία στιγμή να βρίσκουμε μια λύση. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε απλώς να λέμε άντε επιτέλους ας πούμε ένα ναι στο τέλος θα πρέπει στο μέλλον η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι πιο ουσιαστική και θα πρέπει η Προεδρία του Συμβουλίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ουγγρική, Πολωνική, Δανική και Κυπριακή Προεδρία, πιστεύω ότι έχουν απόλυτη συμφωνία μαζί μας για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ενός πιο τακτικού διαλόγου και να ακολουθηθούν οι πρέπουσες διαδικασίες για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις ε, επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές με μια πραγματική διαπραγμάτευση με το Συμβουλίο. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο τώρα των δημοσιονομικών προοπτικών, θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερα κονδύλια από αυτά τα οποία έχουμε κατά τη διάρκεια των τωρινών, της τωρινής δημοσιονομικής ε, περίοδου. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι κάτι το νομοτελειακό, ότι δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τίποτα, γιατί το βλέπουμε στις διαδικασίες του προϋπολογισμού ότι πολλές φορές τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στους περισσότερους εθνικούς προϋπολογισμούς υπάρχει μια μεγάλη θέληση περιστολής και δημοσιονομικής πειθαρχίας λόγω της ε, χρηματοοικονομικής και της ε, ακολουθήσεως σας ε, οικονομικής κρίσης και φυσικά και του γεγονότος ότι πάρα πολλά κράτη-μέλη βρίσκονται σε κατάσταση υπερχρέωσης και επομένως οι προπολογισμοί αυτών των κρατών μελών θα περνάνε προϋπολογισμοί λιτότητος <clears throat> και εξοικονόμησης. Μετά λοιπόν από το 2013 και δεν είμαστε μακριά, δύο χρόνια απέχουμε, θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να ξανααναφερμάνουμε την οικονομία της Ευρώπης και θα πρέπει να μπορούν και οι προπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξουν κάποιο ρόλο για κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε γαλαντόμες <clears throat> ενέργειες και να δώσουν περισσότερα χρήματα τα οποία ξεπερνούν το τωρινό επίπεδο. Ήδη υπάρχει το, η οροφή αυτή που γνωρίζετε, το 1,23% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οροφή σε σχέση με τις δαπάνες μας. Πιστεύω ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές που θα εξέλθουν από τη διαπραγμάτευση θα πρέπει να βρισκόνται λίγο κάτω από το 1,23% για να έχουμε και κάποιο περιθώριο. Αυτό πάντως το οποίο εμείς επιθυμούμε και μπορείτε να το διαβάσετε και στην έκθεση της Επιτροπής μας, είναι να υπάρχει μια συμφωνία με το Συμβούλιο για την ε, ευελιξία, <clears throat> για την ευκαμψία. Όχι ένα στενός κορσές που θα προέλθει από αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα όταν για οποιοδήποτε λόγο τα κονδύλια του προϋπολογισμού δεν έχουν εκταμιευθεί, εάν χρειάζονται κάπου αλλού, να υπάρχει δυνατότητα με ένα σχετικά απλό τρόπο, με μια εύκαμπτη διαδικασία, τα χρήματα αυτά να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές του προϋπολογισμού. Αυτή είναι η έννοια της ευελιξίας για μας. Τώρα για το πόσα χρήματα θα πρέπει να μπουν σε ποιο πλαίσιο και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια ενδεικτική κατανομή στις διάφορες κατηγορίες του προϋπολογισμού για το θέμα αυτό ακόμα θα πρέπει να συζητήσουμε και στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, δεν έχει τελειώσει η επεξεργασία αυτών των θεμάτων. Έχουμε μερικές ακόμα συνεδριάσεις και ελπίζουμε ότι στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου θα πάρει την τελική της μορφή η έκθεσή μας και στη συνέχεια τον Ιούνιο θα έλθει αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια και για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά και θέλουν να καταθέσουν ενδεχομένως η προθεσμία για τις τροπολογίες στη δική μας Επιτροπή η είναι 31η Μαρτίου. Και όποιος θέλει να κάνει τροπολογίες λοιπόν μέχρι τότε θα πρέπει να κάνει για την Επιτροπή Σούρα θα πρέπει να τις υποβάλει μέχρι τότε. Αν θέλετε μπορώ να κλείσω εδώ. Την Πέμπτη εμείς συνεδριάζουμε και πάλι και το πρωί και το απόγευμα. Και φυσικά όλοι αυτοί και όλες αυτές που ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν διότι είναι ανοιχτέ η θύρε μας. Και το λέω πάντα αυτό σε όλους, σε όλες τις επιτροπές ότι είμαστε μια επιτροπή η οποία είναι έκτακτη επιτροπή, είναι ειδική επιτροπή, αλλά ό,τι ισχύει για τις άλλες επιτροπές ισχύει και για μας. Έχουμε μια έκθεση, ένα σχέδιο από τον εισηγητή, που κατατίθεται μπορούν οι συνάδελφοι να καταθέσουν τροπολογίες. Σε αυτό το σχέδιο συζητούμε αυτές τις τροπολογίες μεταξύ μας και καταλήγουμε εν καιρό <clears throat> σε κάποιες ε, συμβαστικές λύσεις και καταλήγουμε σε μια ψηφοφορία, ενδεχομένως με αντιπαράθεση, στην τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και μετά παραπέμπεται η έκθεση στην Ολομέλη. Αυτή είναι η φυσιολογική διαδικασία επεξεργασίας των εκθέσεων. Αυτό θα κάνουμε και εμείς και εδώ θα κλείσω και περιμένω τις ερωτήσεις που ενδεχομένως θα θέλετε να θέσετε. Να θέσουν οι συνάδελφοι ή οι συνάδελφες, γιατί βλέπω να υπάρχουν μόνο γυναίκες εδώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Χάουκ. Μας ε, παρουσιάσατε ιδιαίτερα πλούσιο υλικό. Και όπως είπατε, αυτά τα θέματα είναι αποφασιστικά για το μέλλον. Είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να μπορέσει σε όλες αυτές τις προκλήσεις να θέσει και την πρόκληση της ισότητας των φύλων. Οι συντονιστές πρότειναν να καταθέσουμε μερικές τροπολογίες και πριν δώσω το το χρονοδιάγραμμα θα ήθελα να μιλήσουν ε, οι συνάδελφοι σχετικά με την έκθεση. Η κυρία Κορνέλησεν. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας δείτε. Κυρία Χάουγκ, λέει η κυρία Κορνέλησεν. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εισαγωγή και η εισήγηση. Αλλά έχω μια-δυο παρατηρήσεις ή και ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ μαζί σας και με το παραπάνω όσον αφορά την έμφαση που να δοθεί στην υπόθεση πολιτική 2020 και να υπάρξει ένας προϋπολογισμός της Ένωσης. Όλοι οι προβλησμοί τέλος πάντων να αναφυγραμμίζονται για να μπορέσει κάτι να βγει από την υπόθεση. Και επίση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι ή στην έκθεση ή στο ε, σχέδιο έκθεση παιδάκι Αναγνωρίζετε το τι προκλήσει και αντιμετωπίζει η κοινωνία για τα μέσα επόμενα χρόνια. Όμως, η γυναική υπόθεση δεν την υπόψη καθόλου. τα θέματα των δύο φίλων. Και τελικά, οι δυνατότητες που δίνονται όσον αφορά αυτούς που έχουν το πρόβλημα. Δηλαδή, τις γυναίκες εργαζόμενες. Για πέστε μας τώρα. Η, Επιτροπή σας κάνει τίποτε για να εκπαιδεύσει τα μέλη της όσον αφορά τον προπολογισμό αναφύλλω. Γιατί πρόσφατα έχουμε κάποιες μελέτες για τον κοινωνικό προπολογισμό και πώς λαμβάνει ή δεν λαμβάνει υπόψη τους άρενες ή φίλες Ευρωπαίους. Μήπω Μήπως πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής σας πάνω σε αυτό. Επίσης, για πέστε μας. Τι θα κάνετε αφού παρουσιάσει ό,τι θέλει να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, πότε κατάλαβα, Υπάρχει θέμα το κατά πόσον όταν προσφέρει τι προτάσει στην Επιτροπή, αν ακόμα θα λειτουργεί η δική σα Επιτροπή. Τι θα κάνετε. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλη, είναι η κυρία Τόμψον. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάουγκ. τόσο μας εξηγήσατε έχουν βαθιά νοήματα όσον αφορά τις δημοσιονομικές προτάσεις. Όντως είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το ότι κατά τι ισότητας των ευφύλων δεν λαμβάνεται υπόψη πρώτα Επιτροπής. Θα καταβάλουμε εμείς προσπάθεια. Αλλά είναι πολύ παράδοξο ότι δεν λένε τίποτα και όταν μιλάμε για τον γεράσκοντα πληθυσμό, γνωρίζουμε ότι το 2025 το 10% των Ευρωπαίων πρόκειται να είναι 85 ή μεγαλύτεροι. Και 90% αυτών θα είναι γυναίκες. Τώρα, όσον αφορά την ε, έκθεση έχουμε ξεκαθαρίσει τα στοιχεία που υπάρχουν. Ότι υπάρχουν πάρα πολλέ σοβαρέ μισθολογικέ διαφορέ και διαφορέ στι συντάξει. Μιλάμε για 50%, 75,5%. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να αποτυπωθούν στο κείμενο. Το συζητήσαμε και το ψηφίσαμε το κείμενο μας τον ε, Δεκέμβριο όσον αφορά το δουλεμπόριο ανθρωπίων όντων, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα. Μας ικανοποιεί πάρα πολύ σχετική οδηγία. Το πρόβλημα αυτό όλο ένα και εντείνεται. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στις προσπαθίες τους κατά αυτού του εμπόριου λευκής αρκός, γιατί από ό,τι φαίνεται τα κράτη-μέλη δεν έχουν αρκετούς πόρους. Ιδίως όταν υποδέχονται πάλι τις γυναίκες που επαναπατρίζονται, που έχουν περάσει αυτά τα δίνα Και στη Βουλγαρία μας τα εξήγησαν που πήγαμε. Τέλος. Έχω ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει σχέση με τα δύο φύλλα αλλά διακρίνω σε αυτή την ε, πρόταση ότι θέλετε να μείνουν στα ίδια επίπεδα και ταυτόχρονα λέτε όμως ότι θέλετε να αυξήσετε τον προβλημα για την έρευνα. Πώς θα γίνει αυτό, πού θα πάρετε τα χρήματα, μήπως θα πάρετε από τα διαστοτικά ταμεία. Διότι έχουν δραστηριότητα τέτοια όσον αφορά την ανεργία ε, στις ομορφισμένες περιοχές, κάτι που είναι πολύ ανεργια στις ομορφισμενες περιοχες κατι ειναι πολυ σημαντικο για τη η υπόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Παρβάνοβα, και εγώ κυρία Πρόεδρε, έχω μια-δυο ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα, ναι θα πρέπει να βάλει υπόψη τις διαφορές των δύο φύλων, ο προπολογισμό. Επίσης να καλύπτονται και οι πιο ευάλωτες στο δημοσιογραφικό οι γυναίκες δηλαδή, αλλά και θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό το οποίο ήδη συζητήσαμε εδώ, δηλαδή φτώχεια, εθνικές μειονότητες. Πολύ σημαντικό αυτό. Και το κοινωνικό ταμείο επίσης θα πρέπει να καλύψει περισσότερο τις φτώχε γυναίκες. Κάτι γνώμη μου. Υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο ε, κάποιες πρακτικές όπως στην Ισπανία που είναι παράδειγμα προς για αυτό το πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο και να δούμε κατά πόσο αυτά μπορεί να τα μεταφέρουμε στο κοινωτικό επίπεδο. Και επίσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για τον κοινωτικό προπολογισμό. Ευχαριστώ κυρία Παπανούβα. Η Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Χάουγκ, να παρουσιάσετε τη δουλειά σας στην Επιτροπή Γυναικών. Εδώ, εδώ είμαι. Όσο μόνιμη εισηγήτρια για το θέμα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Μιλάτε εσείς ε, για τις ε, προκλήσεις κλειδί ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μια κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση και στην κατάρτιση. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να τονίσετε την προβληματική των γυναικών στη διαβίου κατάρτιση και τις δυνατότητες που θα πρέπει να δώσουμε στις γυναίκες για να κρατήσουν τη δουλειά τους ή για να επανέλθουν στον εργασιακό βίο. Ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα ευπαθής πληθυσμός ε, οι γυναίκες. Και το να καταβάλουν προσπάθειες για κατάρτιση μαζί με τη δουλειά και την οικογένεια είναι πολύ πιο σκληρό για τις γυναίκες. Θα ήθελα να έχουμε λοιπόν ειδικέ πολιτικές για τις γυναίκες για να τις υποστηρίξουμε στην απασχόληση στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το εξετάσουμε συλλογικά. Πρέπει να επιδείξουμε μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ για αυτήν την ενδιαφέρουσα εισαγωγή. Φαντάζομαι ότι η Επιτροπή μας θα τα λάβει υπόψη της όλα αυτά και θα τα συμπεριλάβει στην προβληματική της. Αν κατάλαβα καλά, στην έκθεσή σας υπογραμμίζεται δύο πράγματα, αφενός τις προκλήσεις κλειδί, την δημογραφική πρόκληση και την ενεργειακή πρόκληση, όπως επίσης και τη διαπίστωση ότι χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και ότι η Ευρώπη μπορεί να συνεισφέρει με προστιθέμενη αξία στην επίλυση της κρίσης. Πρόκειται για, μια, για ένα ζήτημα που είναι εγκάρσιο σε πολλές από τις αποφάσεις μας να βρούμε νέες ε, λύσεις, ε, καινοτομίε για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκπληρώσουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020 και πιο συγκεκριμένα ε, αναφέρομαι στην καινοτομία και στην απασχόληση. Θα έπρεπε Φαντάζομαι να έχουμε τα ευρωμόλογα ή άλλες μορφές χρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ελπίζω ότι θα τα προθίσετε όλα αυτά. Και πολλές διεθνείς μελέτες λένε ότι υπάρχει ο παράγοντας W, γυναίκες στα αγγλικά. που μπορεί να αποτελέσει πρόσθετη αξία. Εμείς όταν μιλάμε για απασχόληση σήμερα αναφερόμαστε κυρίως σε γυναίκες, νέες γυναίκες και για να μπορέσουμε <coughs> να απασχοληθούν αυτές οι γυναίκες δεν αρκεί το να λέμε το 75% και να θέτουμε αριθμητικούς όρους. Πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο. Απασχόληση χωρίς εκμετάλλευση σίγουρα, τα skills, αλλά και καινοτομία στο welfare που δεν είναι κόστος, αλλά είναι επένδυση. Και κάτι άλλο που μπορεί να φανεί περίεργο, να κάνετε μία ανοίξη στην εγκληματικότητα. Σήμερα έχουμε στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας, και στην απασχόληση επίσης λόγω της εγκληματικότητας, δηλαδή η εγκληματικότητα αφαιρεί καθαρούς πόρους, δημόσιους πόρους, επηρεάζει την πραγματική οικονομία των χωρών, όχι μόνο στην Νότια Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Και τελευταίο σημείο θα ήθελα να καταλάβω για τους νέους. Οι νέοι λέτε το 2020 μετά από την σχολική πανεπιστημιακή τους εμπειρία θα πρέπει να έχουν εγγύησεις και αυτό σήμερα δεν τον γιάται κανείς. Πρέπει να γίνει μια πλήρης αντιστροφή της προοπτικής ε, του προϋπολογισμού για να αλλάξει και η στρατηγική οπτική στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Κώστα. Η κυρία Λούλινγκ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ χρειάστηκε να έρθω από το Λουξεμβούργο και καθυστέρησαμε. Έκανα περισσότερο από μισή ώρες, γι' αυτό καθυστέρησα να έρθω και ζητώ συγγνώμη. Θέλω να θέσω όμως ένα γενικότερο θέμα τώρα. Ο κύριος ε, Λεβαντόφσκι, ο επίτροπος ο οποίος είναι τον προϋπολογισμό, ανέφερε ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι το ποσοστό αύξησης του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το επίπεδο αύξηση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ μίλησα για αυτό το θέμα και στον πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών που μου είπε ότι είναι μη πολιτικά ορθό να αυξάνεται πιο γρήγορα ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπή εν Εγώ δεν νομίζω όμως ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος κρίσης, <clears throat> διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα και άλλες προκλήσεις από ότι η Κομισιόν συγκεκριμένα το θέμα της ε, ε ενδεχομένης εισόδου της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 2012 έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των παρατηρητών, των 18 της Συνδίκης Λισαβόνας. Αν λοιπόν η Κομισιόν δεν θέλει να λάβει υπόψη τα θέματα αυτά, αυτό είναι λαθασμένο για μένα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχει νόημα εδώ να ζητούμε πρόσθετους πόρους για προβλήματα που μας ενδιαφέρουν στην Επιτροπή μας, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα το Κοινοβούλιο να έχει ένα κατάλληλο προπολογισμό. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν την κυρία Χάογκ πώς θα πράξει ώστε η Επιτροπή Προϋπολογισμών να κατανοήσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να έχει υψηλότερο ποσοστό αυξήσεως του προϋπολογισμού του για να καλύψει τις ειδικέ ανάγκες του Κοινοβουλίου. Εγώ ως κοσμήτορ Έχω έρθει σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης στο Λουξεμβούργο και πρέπει να σας πω ότι τώρα θέλουν να μειώσουν τους υπαλλήλους σε διάφορες γλωσσικές μονάδες όταν έχουμε τεράστια προβλήματα για να παίρνουμε εγκαίρως τα κείμενα επί των οποίων θα πρέπει να ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές. Και εμείς έχουμε θεσπίσει τον κανόνα ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα κείμενο εάν δεν υπάρχει σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσει το Κοινοβούλιο εάν δεν έχει εγκαίρως τις μεταφράσεις των κειμένων αυτών και σίγουρα εάν υπάρξει μείωση του αριθμού των μεταφραστών και χαθούν ανθρώπινοι πόροι Εάν το Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να έχει εγκαίρω τα κείμενα τα οποία πρέπει να ψηφίσει, δεν θα μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Θα πάτε λοιπόν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εν ώψη όλων αυτών των στοιχείων να τους εξηγήσετε ότι δεν έχει τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας η Κομισιόν και τους ίδιους περιορισμούς. Όπως ξέρετε θα έρθουν άλλοι 18 συνάδελφοι που αντιστοιχούν στις διάφορες χώρες πέραν του αριθμού των βουλευτών που έχουμε ήδη και πέραν των <clears throat> επερχομένων Κροατών συναδέλφων. Άλλοι 30 βουλευτές λοιπόν θα έρθουν. Μα δεν μπορούμε να παραμείνουμε κάτω από τις συνθήκες στο ίδιο ποσοστό αύξηση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου, βλέποντας πόσο μεγάλες είναι οι πρόσθετες ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν. Οι κοινοβουλευτικοί ήδη έχουν προβλήματα χώρου, Ευτυχώς έχουμε κάποια λεφτά στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε τη γραμματεία μας, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε χώρο, γραφεία για να εγκατασταθούν και οι βουλευτές, οι νέοι και οι συνεργάτες. Και πολλές φορές οι αντιπρόεδροι, οι κοσμήτορες, οι επικεφαλής επιτροπών έχουν πιο μεγάλα γραφεία, αλλά οι άλλοι όχι και στο Στρασβούργο στριμώχνονται και δεν μπορούν να χωρέσουν τους συνεργάτες τους. Μα υπάρχει και εργασιακό δίκαιο σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού μας. Θα ήθελα λοιπόν να θίξω αυτά τα θέματα, τα γενικότερα θέματα γιατί είναι απαραίτητο να υπάρξει και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών σε σχέση με τη λήψη των αποφάσεων που επιβάλλονται, είτε υπάρχει κρίση είτε δεν υπάρχει κρίση, χρειαζόμαστε πιο πολλούς υπαλλήλους και πιο πολύ χώρο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λειτουργήσει σωστά. Και εγώ θα ήθελα να ξέρω αν αυτή είναι και η άποψη <clears throat> της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στο ίδιο επίπεδο αύξηση του προϋπολογισμού της Κομισιόν ή αν θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ κυρία Λούλινγκ. Ήταν πολλά τα ενδιαφέροντα αυτά ερωτήματα. Έχουμε πολύ υλικό, το θέμα είναι ευρύ και τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον. Σημαντικότητες οι ερωτήσεις ε, για την προοπτική της ισότητας των φύλων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας αυτή την προοπτική αν θέλουμε να δράξουμε επιτυχώς τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η κυρία Σενκλέχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω πού νομίζω ότι θα τα βρει αυτά τα χρήματα. έχουν 36% αύξηση για τα διπορικά και αύξηση πάλι μεγάλη επίση για τη διασκέδαση αυτή τη σαμπάνια. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά, αφού βλέπετε ότι παντού έχει λιτότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι να βρούμε τρόπους να περιστήλουμε τον προϋπολογισμό μας, όχι να αυξήσουμε τις δαπάνες. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάουκ τώρα έχει το λόγο για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ξεκινήσω από το τέλος. Γιατί εγώ ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και όχι απλώς ως πρόεδρος της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ πρέπει να δώσω μια απάντηση για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του χρόνου. Είναι γεγονός, όπως είπε η Astrid Λούλινγκ, ότι ο κύριος Λεβαντόφσκι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα τα προσκάλεσε με μια επιστολή να μην έχουν μια αύξηση του προπολογισμού τους υπέρτερη του 1 του 100. Αλλά αυτό είναι ήδη παρελθόν πιστεύω. Γιατί και η Επιτροπή Προϋπολογισμών αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα στον προϋπολογισμό ψηφίσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό. Και το Κοινοβούλιο καθόρισε ότι η αύξηση του προϋπολογισμού μας θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο του πληθωρισμού, δηλαδή 2,3%. Αυτό το 1% λοιπόν που προέτεινε ο Γιάννος Λεβαντόφσκι δεν έχει γίνει δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πούμε επιπλέον ότι ο εισηγητής για το λεγόμενο μικρό προπολογισμό, δηλαδή τα άλλα όργανα εκτός από την ε, Κομισιόν, είναι ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντης, ο οποίος είναι και συνάδελφος της κυρίας Λούλινγκ από το ίδιο πολιτικό κόμμα και νομίζω ότι αυτά τα θέματα μπορείτε να τα ξεκαθαρίσετε μαζί του, κυρία Λούριν. Και εμείς <clears throat> ήδη, εν έχουμε αποφασίσει ότι η αύξηση του προπολογισμού θα είναι μεγαλύτερη από, 2, από 1%, θα είναι 2,3% περίπου. Αυτό το οποίο δεν αποφασίσαμε είναι αν θα παραμείνουμε στα πλαίσια της καταρχήν προταθήσας αύξησης, η οποία ήταν περίπου στο 5 0,6% είπαμε ότι πρέπει η αύξηση να είναι σύμμορφη με τον πληθωρισμό. Αυτά σας τα λέω σαν ε, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και όχι ως πρόεδρος της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Και βέβαια ακούσαμε και την κυρία Σίνκλερ η οποία είπε ακριβώς τα αντίθετα από την κυρία ε, Λούλιν και ξέρουμε ότι και μέσα στο δικό μας κοινοβούλιο υπάρχουν αντιμαχόμενες απόψεις για τα θέματα αυτά και πολλές φορές θα πρέπει οι διαφωνίες αυτές να αποφασιστούν με ψηφοφορίες όπου η πλειοψηφία θα λάβει την τελική απόφαση. Επανέρχομαι λοιπόν στα χωράφια της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ που είναι και η αιτία της παρουσίας μου εδώ σήμερα για την κυρία Κορνέλσεν η Επιτροπή μας έχει μία περιορισμένη χρονική διάρκεια. Λέει η εντολή μας ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε την λήψη αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, τις επόμενες, για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Αν το καταφέρουμε αυτό μέχρι τον Ιούνιο να δώσουμε εμεί μία έκθεση, τότε έχουμε εκπληρώσει την εντολή μας και η Επιτροπή μας δεν θα υπάρχει πλέον. Δεν είναι η πρόθεσή μας να ζητήσουμε μια εντολή η οποία θα, είναι, η οποία θα έχει επεκταθεί. Θέλουμε να τελειώσουμε τη δουλειά μας τον ε, Ιούνιο. Τώρα τα θέματα το διαπραγματεύσαμε το Συμβούλιο για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Αυτά είναι θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Φυσικά εγώ συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά όχι σαν πρόεδρος της Επιτροπής Σούρε. Η Επιτροπή Σούρε ελπίζω ότι θα περατώσει τον Ιούνιο την εντολή της και θα πάψει να υπάρχει. <clears throat> Διάσταση του φίλου. Έχετε δίκιο. Αν θέλουμε εμείς να θέσουμε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να εμφανιστεί ως μια γενική διεκδίκηση και τότε η έννοια του mainstreaming χρειάζεται και κάποιο φρεσκάρισμα. Αν δούμε εδώ την έκθεση την οποία έχουμε υποβάλει και ακόμα και τις τροπολογίες οι οποίες έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφής γενική γραμμή. Δεν είναι τα προγράμματα τα οποία θα αποφασιστούν εδώ. Στην έκθεση αυτή τον Ιούνιο εμείς θα αποφασίσουμε ποια είναι η γενική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα πρέπει η Κομισιόν να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες θα έχουν αριθμητικά στοιχεία, τίτλους, επικεφαλίδες και τότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αν εμείς περατώσουμε επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, τότε το θέμα είναι οι πολιτικές οι οποίες θα συμφωνηθούν με το Συμβούλιο να μπορούν να λάβουν σάρκα και οστά με νομοθετικές προτάσεις. <clears throat> Έτσι γίνεται πάντα. Δηλαδή θα έρθει η Κομισιόν, θα μας υποβάλει προτάσεις, τι θα γίνει με το, με το Ταμείο Συνοχής, τι θα γίνει με την αγροτική πολιτική, τι θα γίνει με το τότε 7ο και τώρα το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα Όλα αυτά λοιπόν τα πολιετή προγράμματα θα τύχουν προτάσεων της Κομισιόν και τότε στην πράξη θα πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι και να κάνουμε όλα αυτά τα απαραίτητα να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου. Αλλά εγώ πιστεύω παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. <clears throat> Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα αρνηθεί ακόμα και η Κομισιόν. Γιατί η Κομισιόν και στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει τονίσει πάντα ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ευμάρεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να γίνει αυτό πραγματικό, πραγματικότητα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό απασχολησιμότητος των γυναικών. Και για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την απασχολησιμότητα των γυναικών, χρειαζόμαστε να λάβουν χώρα ορισμένε προποθέσει, παραδείγματο χάρη η παιδική φροντίδα να επεκταθεί σε όλα τα κρατη Ξέρω ότι σε χώρες όπως η Γερμανία υπάρχουν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στον τομέα αυτό. Θα πρέπει επίσης, και αυτό είναι προφανές, να βρούμε τον τρόπο να δώσουμε την καλύτερη κατάρτιση στις νέες γυναίκες, να τις υποστηρίξουμε στη διαδικασία εκπαίδευσής τους και θα πρέπει στις ηλικιωμένες γυναίκες οι οποίες αφού μεγαλώσει τα παιδιά τους έχουν μείνει έξω από το χώρο εργασίας. <clears throat> Θα πρέπει να μπορούμε να, τους, να τις ενσωματώσουμε σε ένα πρόγραμμα για διαβίου εκπαίδευση και να τις ξαναφέρουμε στο χώρο της εργασίας. Αλλιώς το ποσοστό αυτό όπως αποσυγχωρησιμότητας δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ πραγματικότητα. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Μέχρι τότε θα πρέπει επίση να πούμε ότι το Ινστιτούτο για τα θέματα των φύλων να έχει τη σωστή χρηματοδότηση για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όλα αυτά λοιπόν θα λάβουν χώρα μετά από τον καθορισμό των δημοσιονομικών προοπτικών. Προηγουμένως δεν θα υπάρξει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση για τα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο κάνουμε πάντα είναι να λέμε στην Κομισιόν και να τις επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δώσει την απαραίτητη προσοχή στα θέματα της ε, διάστασης του φύλου και στα θέματα της ε, απασχόλησης των γυναικών και στις συνθήκες κατά τις οποίες μπορεί να υπάρχει απασχόληση των γυναικών. Το θέμα δεν είναι να απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο, είναι να έχουν θέσει εργασίας οι οποίες θα είναι κάτω από καλές συνθήκες. Και η κυρία Μωρέν έχει απόλυτο δίκιο. Το κοινωνικό ταμείο είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία και αυτό τονίστηκε και στις συζητήσεις μας μέσα στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, το κοινωνικό ταμείο είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στις γυναίκες, όχι μόνο στις γυναίκες φυσικά, αλλά και στις γυναίκες. Και επομένως θα πρέπει να δώσουμε μια απαραίτητη προσοχή και μέρημνα στα θέματα αυτά όταν έρθουμε στο θέμα της ε, νομοθεσίας. Υπάρχει ένα άλλο σημείο το οποίο ίσως να είναι και επίμαχο λένε πολλοί, θεωρούν πολλοί, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με ποσοστώσεις. Εγώ το προτείνω αυτό το πράγμα, ότι όταν φτάσουμε στο επίπεδο της ε, νομοθεσίας θα πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένες ποσοστώσεις. Και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη θα πρέπει και αυτά να συνενέσουν στην εφαρμογή αυτών των ποσοστώσεων. Γιατί όπως ξέρετε ποτέ η χρηματοδότηση των προγραμμάτων δεν είναι 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι εν μέρη ευρωπαϊκές και εν μέρη κρατικές πιστώσεις, εθνικές πιστώσεις, αλλά θα πρέπει εμείς να επιμείνουμε ώστε να μην λησμονηθεί η διάσταση του mainstream σε αυτά τα προγράμματα, γιατί πολύ συχνά έτσι γίνεται. Εγώ ξέρω το δικό μου κράτος ε, μέλος από το οποίο προέρχομαι και ξέρω ότι πολλές φορές και στη χώρα μου και στην ε, και στο κρατήδιό μου έχουμε παραγματικά χάρη οι οποίοι μένουν άνεργοι γιατί κλείνει το, το, το ανθρακοροχείο τους και παίρνουν επιδοτήσεις ενώ οι γυναίκες οι οποίες μένουν άνεργες δεν παίρνουν πεντάρα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν και κάποιες ποσοστώσεις και έχουμε πολύ καλούς λόγους για κάτι τέτοιο, γιατί αν θέλουμε να υπάρξει εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η στρατηγική αυτή εμπεριέχει και ποσοστός και θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε αυτές τις ποσοστώσεις. Και το ερώτημα το οποίο θέσατε για τη χρηματοδότηση, ότι θα πρέπει να τα βγάλουμε πέρα με περίπου τα ίδια χρήματα που έχουμε για την αγροτική πολιτική, θα πρέπει να έχουμε τα ίδια χρήματα για την ε, πολιτική <clears throat> συνοχής. Από πού θα βγάλουμε τώρα τα λεφτά για να φτάσουμε το στόχο της ε, έρευνας και ανάπτυξης 30% παραδείγματος χάρη για άλλες πολιτικές. Για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση εδώ. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει μια λύση για τα θέματα αυτά και θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε κάποια σενάρια τα οποία θα εκπονήσουμε και να πούμε στο Συμβούλιο αν δεν θέλετε το Α ή το Β, τότε αυτή η πολιτική δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να την επομισθούν τα κράτη-μέλη και μόνο. Και όταν σας λέω για τάξη μεγέθους, <clears throat> αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ακριβώς τα ίδια χρήματα. Σας λέω ότι έχουμε την ίδια τάξη μεγέθους και στην επόμενη περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σημαντικά μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Έχουμε τώρα περίπου 1,2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι πολύ περισσότερο. μπορεί να έχουμε μια χρηματοδότηση της τάξης του 1,04, 1,06. Εξαρτάται λοιπόν από την ε, διαδικασία χρηματοδότησης ενός ε, προγράμματος, το οποίο μπορεί να χρειάζεται πολλά χρήματα εκκίνησης, μετά να υπάρχει μια κοιλιά και μετά πάλι χρήματα στο τέλος. Αλλά αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε σε συγκεκριμένο επίπεδο. Το άλλο το οποίο θέλουμε επίσης είναι να υπάρξει ενισχύση και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανασυγκρότησης, για την Ανατολική Ευρώπη δηλαδή, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε και οι δύο τράπεζες με τις ενεργειές τους να ενισχύσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι θα προσελκυστεί και το χρήμα του δημόσιου τομέα από τα κράτη-μέλη και πολλές φορές να, αντιμε, να αντικατασταθούν πιστώσεις οι οποίες δεν μπορούν να δοθούν από τα κράτη-μέλη. Όχι μόνο να αντικαταστήσει λοιπόν την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την εθνική χρηματοδότηση και να υπάρξει και μια κοινή αντιμετώπιση από τις τράπεζες αυτές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω συζητήστε και με τους συναδέλφους σας και τις συναδέλφους σας στα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί και αυτές θα πρέπει να μας υποστηρίξουν και να ασκήσουν πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν ξέρω αν τα έχω καλύψει όλα τα ερωτήματα τα οποία μου θέσατε. Νομίζω σε γενικές γραμμές ναι, το έχω πράξει. Όπως σας είπα λοιπόν, η διάσταση του φίλου είναι πράγματι αυτό θα το τονίσουμε <clears throat> σε επίπεδο γενικό, ίσως με ένα ε, ιδιαίτερο κεφάλαιο και να πούμε ότι όταν έρθουμε στις νομοθετικές προτάσεις δεν θα πρέπει να λησμονηθεί αυτό το gender budgeting, η εγγραφή δηλαδή στο προπολογισμό επιβάση φύλου. Ευχαριστώ κύριε Χάουκ. Η Επιτροπή μας θα καταθέσει τροπολογίες και έτσι θα, θα προσπαθήσουμε κι εμείς προοπτική της ισότητας των φύλων να είναι παρούσα στην έκθεση της ε, ΣΟΥΡΕ και να παραμείνει και σε όλες ε, τις ε, εργασίες του προπολογισμού. 28 Μαρτίου στις 12 λίγη προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Στις 20 Απριλίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην ε, Σούρε θα ψηφίσουν στα τέλη Μαΐου. Η έκθεση θα περάσει τον Ιούλιο από την ε, Ολομέλεια. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την κυρία Χάουγ για την παρουσία της. κυρία Χάουγ. Κάτι ακόμα, ένα ερώτημα μάλλον το οποίο πρέπει να σας θέσω. 31 Μαρτίου, όπως σας είπα, είναι καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες. Αν η Επιτροπή σας, οι μεμονωμένες συνάδελφοι από την Επιτροπή σας θέλουν να καταθέσουν τροπολογίες, πρέπει αυτό να γίνει μέχρι τις 31 ε, Μαρτίου. Αλλιώς δεν μπορούμε να τις επεξεργαστούμε τις τροπολογίες αυτές. Ακόμα και αν μια επιτροπή κάνει τροπολογίες, αυτές δεν θα πάνε αυτόματα στην Ολομέλεια, θα πρέπει να περάσουν από ψηφοφορίες μας. Ναι, ίσως να υπάρχει μια παρεξήγηση. Εμείς θα καταθέσουμε τις τροπολογίες. Θα τις ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και μετά θα έρθουν στο κείμενο της Σούρε. Δεν είναι τροπολογίες επί του κειμένου της Σούρε, είναι οι τροπολογίες στη δική μας έκθεση. Θα ψηφίσουμε λοιπόν κατευθείαν εμείς τις τροπολογίες μας. Σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια των εργασιών. Πάμε στο σημείο 5. Η δημογραφική αλλαγή και οι συνέπειές της για τη μελλοντική πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη στο παρελθόν ε, συζητήσαμε για τις ε, δημογραφικές αλλαγές και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους. Έχουμε μία εισηγήτρια, την Άννα Ζαμπόρσκα. Και αυτή η γνώμη θα κατατεθεί στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων που είναι και αρμόδια επί της ουσίας. Δίνω το λόγο στην κυρία Ζαμπόρσκα για να μας πει πώς οργανώνει τις εργασίες της. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, μάλλον ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση και νομίζω ότι η πολιτική της συνοχής μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά τα, τα δημογραφικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Όπως προείπα και όπως είπατε για σωστά κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή μας έχει συζητήσει ήδη από το 2006 το πρόγραμμα αυτό. Και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δημοσιεύσει την πράσινη βίβλο που αφορούσε τα δημογραφικά και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Έχουμε μετά και εμείς εκπονήσεις στη συνέχεια μια σειρά εκθέσεων. Και νομίζω ότι μπορούμε να το εντοπίσουμε και τον χαμηλό αριθμό και ρυθμό γεννήσεων αλλά και την γύρανση του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η πολιτική συνοχής είναι δυνατόν επομένως να βελτιώσει την κατάσταση να επηρεάσει θετικά των των γεννήσεων αυτό μπορεί να γίνει με τις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας και προνοίας και επίσης να φροντίσει αυτούς οι οποίοι ε, βρίσκονται σχεδόν στην ηλικία συνταξιοδότησης που μπορεί να τους βοηθήσει να βρουν κάποια απασχόληση. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με τα επιμέρους ζητήματα του δημογραφικού ελλείμματος. Ήδη έχω κατεβάσει κάποιες προτάσεις για το πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση, ιδίως δε κάποιες προτάσεις που αφορούν τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές. Η ευθύνη των περιφερειών ε, και αρμοδιότητες είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα μέλος και τα πράγματα εξαρτώνται επομένως από το τι αρμοδιότητες έχουν αυτές οι περιφέρειες. Πάντως δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή της επικουρικότητας και θα πρέπει επίσης να αξιοποιούμε και τις περιφερειακές πολιτικές εκείνες οι οποίες σχετίζονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάρα πολύ ενδιαφέρον προσθέσει στο θέμα, διότι έχουμε κάποιες περιφέρειες οι οποίες είναι πιο κοντά στον κόσμο. Και νομίζω ότι στην εκθεσή μου θα ασχοληθώ συγκεκριμένα με κάποια συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία ε, έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχή και ταυτόχρονα με τη γυναική υπόθεση, το γυναικείο ζήτημα. Διότι στα μια καθημερινή, αλλά βέβαια και στην Ευρώπη των 15 αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο φαινόμενο της φυγής εγκεφάλου. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ήπεθρο. Και την αναστηφιλία. Πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό. Επίση, θα πρέπει να δούμε πώ θα τονώσουμε την απασχόληση στην Ήπεθρο. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα και επομένω να σταματήσουμε αυτή την φυγή των νέων γυναικών, οι οποίε πολύ συχνά το κάνουν αυτό, πρώτα έχουν ένα σωρό δεξιότητε, πρώτα ότι είναι μορφωμένε. Υπάρχει τώρα και κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε επανειλημμένα. για το πώ θα γίνει συμφιλίωση, συγκερασμό, συνδυασμό επιτυχία τη επαγγελματική με την ε, οικογενειακή ζωή. Επομένω και αυτό θα βοηθήσει όσον αφορά τον ρυθμό των γεννήσεων και θα βοηθήσει στην πλαισίωση και φροντίδα των ε, πιο ηλικιωμένων. Μην ξεχνούμε τι είναι με τις φτωχές γυναίκες, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η φτώχεια χτυπάει κατεξοχήν τις γυναίκε ενημέρωση, μικροχρηματοδότηση, νέε τεχνολογίε, όλα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις γυναίκε αυτέ στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής, ε, όπου αυτά τα προβλήματα σοβούν στην Ευρώπη ή αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αυτή η μελέτη του ΩΣΑ ε, αυτό έγινε με την ευκαιρία της μέρας της γυναίκας και είπαμε ότι 30 με 40% της ε, λεγόμενης αόρατης εργασίας, αφανούς εργασίας, γίνεται από γυναίκες. ότι θα έπρεπε η Eurostat στα στατιστικά της δεδομένα να καλύψει και αυτές τις μεταβλητές και αυτά τα στοιχεία. Αυτή την εργασία που είναι αφανής και δεν αμείβεται και κυρίως ασκείται από τις γυναίκες. Επίσης έχουμε και ε, την ασχόληση των γυναικών με ε, εθελοντική δραστηριότητα. Ελπίζω ότι η Eurostat πρόκειται να ε, επεξεργαστεί τους σχετικούς δείκτες, ούτως ώστε να μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο βαθμό οι γυναίκες ασχολούνται με τέτοιες εθελοντικές δραστηριότητες <coughs> Μιλούμε για τη γύρανση του πληθυσμού και ξέρουμε ότι το 2012 θα είναι το, η χρονιά ε, των ενεργών γυρατιών. Οπότε, γι' αυτό και εγώ θα ασχοληθώ με την δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι Και επίσης να δούμε το πώς η κοινωνική και η περιφερειακή συνοχή θα βελτιωθεί. Έχουμε κάποιες περιφέρειες που είναι πιο φτωχέ από άλλε. Να δούμε επομένω πώ θα υπάρχει καλύτερη αυτών των δραστηριοτήτων για αυτέ τι ευάλωτε περιοχέ. Να χρησιμοποιήσουμε το περιφερειακό ταμείο ενδεχομένω. Και επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω τι γίνεται με την δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες σε μια τέτοια συγκυρία κρίσης. Υπάρχει πρόβλημα με την απασχόληση και αυτό το τονίζω στην εκθεσή μου. Άρα, να ασχοληθούμε για το πρόβλημα της απασχόλησης αυτών των πιο ηλικιωμένων γυναικών και επίσης υπάρχουν διάφορες πολιτικές που ασχολούνται με αυτές τις ε, γυναίκες σε σχέση και με την οικογενειακή ζωή. Χρειάζεται επομένω να έχουμε μια φρέσκια, μια καινούργια, νεοτεριστική ματιά στο πρόβλημα αυτή την έκθεση. Και να δούμε πώς μπορεί ο ρόλος της γυναίκας να πλησιωθεί καλύτερα. Πρώτα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο να παρουσιάσω το κείμενό μου και είμαι σίγουρη ότι οι συνάδελφοι θα προχωρήσουν σε διατύπωση τροπολογιών, σχολείων, ερωτήσεων. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρσκα. Δίνω το λόγο στην Αντιπρόεδρό μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να εγκομιάσω την εργασία της κυρίας Ζαμπόρσκα. Η ανάλυση της είναι πάρα πολύ καλή. Για τους στόχους υπάρχει ένα σημείο που θα ήθελα να δούμε, είναι το σημείο 6. Σε αυτό το σημείο Ζητάτε ο Ουροστάτ να διαμορφώσει δείκτες για τη συμμετοχή των γυναικών στην εθελοντική εργασία. Εγώ θα ήθελα όμως αυτό να το τραβήξουμε κάπως παραπάνω. Επειδή ο στόχος είναι να, να αξιολογήσουμε την γυναικεία δουλειά, θα έπρεπε πέρα από το αίτημα προς την Οροστάτ μαζί με περιφερειακές αρχές να κάνουμε μία αξιολόγηση των κεκτημένων ικανοτήτων. Αυτή η εθελοντική εργασία θα πρέπει να επιτρέπει στις γυναίκες με μία αναγνώριση ικανοτήτων να οδηγηθούν στην αμοιβόμενη εργασία όπως οποιοδήποτε, οποιοδήποτε άλλος που θα είχε την ε, δυνατότητα να έχει μία πιο ακαδημαϊκή κατάρτιση. Αν θέλουμε να είμαστε πιο ε, ριζικοί κυρία Ζαμπόσκα, θα πρέπει να τονίσουμε αυτήν την δυνατότητα για τις γυναίκες. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Λέει η κυρία Μπάουερ, είναι πολύ ενδιαφέρον που γύρεται το θέμα αυτό υπό την έποψη της πολιτικής συνοχής από τη μία πλευρά και της δημογραφικής αλλαγής από την άλλη πλευρά εστιάζοντας στην κατάσταση των γυναικών. Είναι πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση και πιστεύω ότι το σημείο εστίασης είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον. Για τους λόγους αυτούς πιστεύω ότι το θέμα της υποδομής στην πολιτική συνοχής είναι ένα κομβικό θέμα. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαι πεπισμένη ότι μπορεί να είναι κάπως μονομερής η παρουσίαση στη γνωμοδότηση αυτή του θέματος γιατί εδώ δεν εμπλέκεται μονάχα το θέμα της κοινωνικής υποδομής. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για την ολιστική προσέγγιση της κυρίας Ζαμπόσκα. Ίσως θα ήταν χρήσιμο βέβαια να θέσουμε ευρύτερα το θέμα των υποδομών και της πολιτικής συνοχής και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της θέσης των γυναικών στη διαδικασία αυτή για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση το να δημιουργήσουμε μια προσθέμενη αξία στα θέματα αυτά, αλλά πιστεύω επιπλέον ότι αξίζει να εργαστούμε στον τομέα αυτό, γιατί η μελλοντική πολιτική συνοχή μπορεί να παίξει ένα κομβικό ρόλο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Eh, eh, η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ την Άννα Γαβρόσκα για, την, για τις ε, προτάσεις της, είναι ιδιαίτερα εύστοχες. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να βρούμε ποια είναι τα κεντρικά του σημεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να τολίσουμε τις περιφερειακές πολιτικές κυρίως αυτή τη φάση μεταρρύθμισης των στόχων των περιφερειακών πολιτικών. Το θέμα της ε, αόρατης εργασίας ήταν και μια έκκληση που απευθύνθηκε στο Πεκίνο, στη διάσκεψη του Πεκίνου, να μιλήσουμε για την οικονομική και κοινωνική αξία του έργου της φροντίδας, το οποίο δεν παράγει μεν πλούτο, αλλά παράγει αξίες. Αυτό το είχε ζητήσει και ο ΙΕ να γίνει μία μέτρηση. Όταν μιλάμε για μικροπίστοση, θα πρέπει, όχι μόνο για την εμπορική δραστηριότητα, στα Ιταλικά λέει commerciale, εμπορική δυνατότητα, trade θα έπρεπε να πούμε στα Αγγλικά, για να μπορέσουμε να μειώσουμε την φτώχεια των γυναικών μέσω των μικροδανείων. Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι να εγγυθούμε τη μεγαλύτερη αυτονομία των ηλικιωμένων. Και αυτό μέσα ε, να μπορέσουμε να εγγυθούμε την αυτονομία σε περιφερειακό επίπεδο οργανώντας το σύστημα των βάουτσερ, των, κουπουνιών για τη φροντίδα κατοίκων των ηλικιωμένων. Πρόθεση επίσης των ανθρώπων τρίτης ηλικίας ενισχύοντας τα δίκτυα εκείνα που τους βοηθούν ας πούμε στην Ιταλία έχουμε το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας θα πρέπει δηλαδή να ενισχύσουμε αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι εργάζονται μεταξύ των, για, για, για, τη σχέση μεταξύ των γενεών για παράδειγμα την κατάρτιση στην πληροφορική Επίσης, ε, την βοήθεια στην οικογένεια για τη βοήθεια της αυτονομίας του ηλικιωμένου. Είναι πράγματα που απασχολούν ιδιαίτερα τις ε, περιφέρειες. Εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κύριος Ρόλαντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λίγα λόγια. Προς πληροφόρηση. Τέλη Μαρτίου θα παρουσιάσει η Κομισιόν για την έκθεση για την ε, δημογραφία. Πρόκειται για μια, διετή, μια, για μια έκθεση που ε, εκπονείται κάθε δύο χρόνια. Έπρεπε να είχε δημοσιευθεί πέρυσι, θα δημοσιευθεί τώρα. Έχουμε καλά νέα για το ποσοστό γονιμότητας και γεννήσεων ποσοστά τα οποία συνδέονται και με την εργασία των γυναικών αναλογικά πρόκειται για μία μικροσυνοχή δηλαδή οι πολιτικές ενισχύονται προς τη σωστή κατεύθυνση τώρα για την ε, για την φυγή των εγκεφάλων διαπιστώνουμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ένα αρνητικό υπόλοιπο στη μετανάστευση έχουν περάσει σε θετικό πλέον επίπεδο. Αυτό είναι καλό για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Για το σημείο 7 Θα αναφέρω στους ε, συναδέλφους μου που είναι επιφορτισμένοι με το ευρωπαϊκό έτος να αναλάβουν αυτά τα ειδικά μέτρα για τις γυναίκες και να μην τις ξεχάσουμε τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν θέλετε άλλα στοιχεία, είμαι στη διάθεσή σας. Κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ και όλους τους ε, συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Να σας πω. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι προτάσεις θα καλυφθούν από την τελική εκδοχή του κειμένου μου και σας ε, ευχαριστώ για όλα όσα είπατε, που σίγουρα θα συμβάλλουν. Και ελπίζουμε να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. και να σταματήσει και η φιλία στις πιο προβληματικές περιφέρειες, να σταματήσει αυτή η φυγή των εγκεφάλων, κάτι το οποίο άμεσα έχει να κάνει με την επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος. για τη μικροχρηματοδότηση στο σημείο 4 που έχει αναφερθεί. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, ε, πώς θα δούμε ευρύτερα το θέμα. Επίσης, τώρα για τις αρμοδιότητες των περιφερειακών ε, αρχών και τις φορολογικές αρμοδιότητες πιο συγκεκριμένα, αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Άρα σε περιφερειακό επίπεδο δεν μπορούμε κάτι να προτείνουμε. Θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο κάτι να γίνει. Και πάλι ευχαριστώ συνάδελφοι για όσα είπατε και τροπολογίες ε, ε, και προτάσει θα, θα αγκαλιάσω στο, στο κείμενό μου. Ευχαριστώ. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Πάρα πολύ σύντομα λέει κυρία Μπάουερ. Θέλω να αναφέρω ότι Υπάρχει ένα πρόβλημα μετάφραση στο σημείο 5 στα Ουγγρικά. Ευχαριστώ που μας υποδείξατε το λάθος. Η 22 Μαρτίου στις 12 η προθεσμία για τις τροπολογίες. Λοιπόν, 26 Μαΐου θα περάσει από την Επιτροπή στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω μία μικροαλλαγή στην ημερήσια διάταξη διότι ήρθε η Φραντσέσκα Μπαλτζάνη που είναι η συγγήτρια για τον προϋπολογισμό του 2012. Προτείνω, αν συμφωνείτε φυσικά, να αντιστρέψουμε τη σειρά των σημείων και να πάμε στον προϋπολογισμό του 2012. Συμφωνείτε? Ωραία. Πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, ήδη το είχαμε αλλάξει δηλαδή. Προϋπολογισμός 2012. Και δίνω το λόγο στην κυρία Μπαλτζάνη, που είναι η εισηγήτρια για, το για τον προϋπολογισμό του 2012. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ για τη συνάντηση. Είναι μια πολύ χρήσιμη συνάντηση για όλη την διαδικασία του προϋπολογισμού που όπως κάθε χρόνο είναι και πολύ ε, μακροχρόνια και ιδιαίτερα σημαντική. Εγώ θα ήθελα στον προϋπολογισμό να εμπλέξω σε μια λεπτή φάση του προϋπολογισμού τις ε, πιο τομεακές επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου. Στο έγγραφο εργασίας ε, και στην πρόταση που υποβάλαμε θέλησα να προτείνω μόνο γενικές μεγάλες προτεραιότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πλαίσιο, την κορνίζα μέσα στην οποία θα συμπεριλάβουμε τον προϋπολογισμό. Το γενικό πλαίσιο λοιπόν η κορνίζα θα πρέπει να είναι η στρατηγική του 2020. Εμείς πάντοτε ψάχνουμε προτεραιότητες ε, στον προϋπολογισμό. Αυτή η χρονιά όμως αλλάζει. Είναι διαφορετική από τις άλλες διότι μέσα από αποφάσεις ε, ε, που πέρασαν με μεγάλη πλειοψηφία ε, ενέκρινε το Κοινοβούλιο για το 2020 και είναι η πρώτη χρονιά όπου ε, το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στην οικονομική governance και θέλει να έχει το λόγο του στους μεγάλους ε, στόχους της Ένωσης, στη στρατηγική 2020 που για να γίνει πραγματική και συγκεκριμένη θα πρέπει να έχει και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Ξεκινώντας από αυτό το γενικό πλαίσιο, χρειάζεται μεγάλη διαβούλευση, ε, συνέργεια ε, μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών προϋπολογισμών. Αυτό είναι το ένα. Και προσπάθησα να στήσω μια πρώτη πρόταση προτεραιοτήτων ε, ουσίας είναι η πρόταση του πρώτου ψηφίσματος και δευτέρου εγγράφου μετά το έγγραφο εργασίας και που θα το παρουσιάσω στην Ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας. Διαπίστωσα ότι ο μεγάλος στόχος που πρέπει να ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο στόχος που πρέπει να προσεγγίσουμε για το 2020, τόσο πιο πολλή δουλειά έχουμε. Ένα στόχος πολύ σημαντικός κυρίως για τις γυναίκες που είναι οι πολίτες της Ένωσης που έχουν δυσκολίες στην Ένωση να βρουν δουλειά και κυρίως ειδικευμένη εργασία. Θα ήθελα αυτό το κομμάτι να είναι ενισχυμένο στην, στον προπολογισμό του 2010. Δουλειά, δουλειά καλύτερης ποιότητας, κατά συνέπεια, κατάρτιση, αύξηση των ικανοτήτων και των γνώσεων του προσώπου. Και ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι οι επενδύσεις που θα μας επιτρέψουν να δώσουμε συγκεκριμένη αξία στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό θα ήθελα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού να μπορέσω να δω ποιες είναι οι προτεραιότητες των τομεακών επιτροπών και καλό όλους τους συναδέλφους να εργαστούν το νωρίτερο δυνατόν για τα θέματα του προϋπολογισμού, να ορίσουν τις πολιτικές προτεραιότητες θεμελιώδεις για να έχουμε μία πρόταση ε, να έχουμε συνέστηση της ε, πρότασης που θέλουμε να υποβάλουμε και στο προσχέδιο και στην εξέταση του προσχεδίου του που θα έρθει τον Απρίλιο. Εγώ θα υποβάλω την πρότασή μου στις αρχές Μαΐου και για τα σχέδια πιλότους ε, και τις ε, προκαταρκτικές φάσεις θα ήθελα να φτιάξω έναν προσωρινό κατάλογο στην, για την ε, Κομισιόν και να το στείλω όσο το δυνατόν νωρίτερα για να έχουμε ένα feedback από την Κομισιόν και να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις προτάσεις εκείνες οι οποίες έχουν πραγματικά την δυνατότητα να προχωρήσουν. Εμείς μετά ως Κοινοβούλιο θα κάνουμε και τις προτάσεις τροπολογίες τους αριθμούς ε, του προϋπολογισμού. ή το αίτημα που έρχομαι να σας υποβάλω είναι ακριβώς αυτό. Να βρούμε ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητες αυτής της, επιτροπή, αυτής της Επιτροπής Ποιες είναι λοιπόν οι προτεραιότητες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σας. Είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η δουλειά. Έχουμε πολύ περιορισμένα περιθώρια. Είμαστε στο τέλος ε, του δημοσιονομικού προγραμματισμού, θα επανακαθοριστούν οι προοπτικές, έχουμε πολύ μικρά περιθώρια οι θετικές προτεραιότητες αλλά και οι αρνητικές προτεραιότητες, προγράμματα δηλαδή που δεν λειτουργήσαν όπως εμείς το περιμέναμε ή που δεν έχουν πλέον την προτεραιότητα που είχαν κάποτε, την είχαν όταν ξεκίνησαν και τώρα μπορεί να μην την έχουν πια. Αυτή η ιεράρχηση ε, προτεραιοτήτων είναι πολύ σημαντική για να φτιάξουμε έναν σωστό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες. Η κυρία Ματέρα είναι η αρμόδια, αλλά δεν είναι εδώ σήμερα. Η κυρία... Χωρίς μικρόφωνο. Εγώ εκπροσωπώ την κυρία Ματέρα που δεν ήρθε εγκαίρως. <coughs> Και ήθελα να σας υποβάλω μερικά σχόλια και ερωτήσεις. Για, εν ώψη του 2012 που θα αφορά την γύρανση του πληθυσμού ε, και εν ώψη του 2020 θα πρέπει να εγγυθούμε εμεί ε, κονδύλια για την καταπολέμηση της στόχιας. Δεδομένου, τώρα, δεδομένης τώρα της οικονομικής ε, κρίσης, εσείς θεωρείτε ότι τα σχέδια πιλότος θα πρέπει να χρηματοδοτούν επαρκώς για να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Το Ίδρυμα της Ζώντας των φίλων χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσει να είναι λειτουργικό και να βοηθήσει και τα εθνικά Ινστιτούτα και τα κράτη-μέλη για να μειώσουμε τις διαφορές φίλων στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Η κυρία Ματέρα ρωτά Δεν θα έπρεπε να υπάρχει συνεχής χρηματοδότηση του, ιδρύ, του Ιδρύματος της Ισότητας των Φύλων, κατά την κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η κυρία Πρόεδρος. Και εγώ έθεσα τον εαυτό μου στον κατάλογο των ομιλητριών, αλλά θα είμαι σύντομη. Αφού κάνω τα ερωτήματα αυτά, λοιπόν, πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι συμφωνώ για τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος για την Ισότητα των Φύλων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κατά τα άλλα, η κυρία Μπαλτσάνη μίλησε για το θέμα της απασχόλησης που είναι η μεγαλύτερη πολιτική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι και εμείς θα πρέπει να θέσουμε στην πρώτη θέση την προτεραιότητα αυτή την απασχόληση αν ο στόχος αυτός θέλουμε να έχει μια πιθανότητα να επιτευχθεί. Στη συνέχεια όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν ένα αμοιβόμενο επάγγελμα. Τότε πρέπει να εκφράσω και τις ανησυχίες μου. Γιατί δεν πρόκειται μονάχα για δυνατότητες απασχόλησης για τις γυναίκες οι οποίες να είναι περισσότερες, αλλά πρέπει να αυξήσουμε και τη δυνατότητα των γυναικών να ζητήσουν και να επιζητήσουν μια τέτοια εργασία. Βλέπουμε στα κράτη μας μέλη ήδη σήμερα πόσο προβληματικά είναι τα πράγματα με την φροντίδα των παιδιών. Υπάρχουν άλλα κοινωνικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να μπορέσουν να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες στην επαγγελματική ζωή. Αν δούμε και τους εθνικούς προϋπολογισμούς για τα ζητήματα αυτά, που είναι πραγματικά προϋπολογισμοί λιτότητος. Ακριβώς αυτές είναι οι κοινωνικές παροχές οι οποίες περικόπτονται από τους προϋπολογισμούς λιτότητος που δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να εργαστούν, να απασχοληθούν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μέσα στα πλαίσια τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι μια από τι μεγαλύτερε προτεραιότητε να διαμορφώσουμε τι προποθέσει για τι γυναίκε να εργαστούν. Εάν φυσικά θέλουμε να επιτύχουμε του στόχου τη Ευρώπη 2020. Και αυτό φυσικά πρέπει να το σκεφτούμε και στα πλαίσια του προπολογισμού του 2012. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος δυστυχώς. Κάποιος άλλος ήθελε να θέσει ένα ερώτημα, η κυρία Κώστα. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, μέθοδο και την ασυνήθιστη ειλικρίνεια της συνάντησής μας με την κυρία Μπαλσάνη η οποία είπε ότι στις ειδικές το ε, τομεακές επιτροπές ε, δίνει προτεραιότητα. Αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Και δεύτερο, ότι θέλει μια σαφή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, στρατηγικών προτεραιοτήτων. Αυτό εντάσσεται και στην λογική του 2020 και μας ευχαριστεί γιατί εμείς ως γυναίκες δώσαμε ε, αυτή την κατεύθυνση. Σημερίζομαι τη στρατηγική προτεραιότητα για τη φτώχεια. Έχουμε και το follow-up για το ευρωπαϊκό έτος, αλλά και την πλατφόρμα για τη φτώχεια. Γνωρίζουμε ότι η φτώχεια είναι κυρίως γυναική. Στον κόσμο το 80% είναι γυναίκες παιδιά. Αυτό συνδέεται φυσικά με τις συνθήκες ζωής των μητέρων. και αυξάνεται αυτή η φτώχεια. Ορισμένες χώρες όπως η δική μου έκαναν σοβαρές περικοπές στον τομέα του welfare, της ευημερίας. Και θα πρέπει κατά συνέπεια να τονίσουμε τη φτώχεια, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και συνέχεια σε ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τις μικροπιστώσεις, τα μικροδάνεια. Θα ήταν σημαντικό κάτι τέτοιο. Δεύτερο, πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στον στόχο του 75% απασχόλησης ε, για τις γυναίκες αν δεν καταφέρουμε να αν καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι η εργασία των γυναικών στον τομέα της ε, φροντίδας είναι, δεν παράγει κόστος. Πρέπει να τονίσουμε την κοινωνική οικονομία με εργασίες ποιότητας για τις γυναίκες και τους νέους. Για το θέμα των skills Εμείς ε, μετά την Λισαβόνα ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για το δικαίωμα της διαβίου κατάρτισης. Αλλά οι επενδύσεις στην ανάπτυξη αυτών των πολιτικών είναι πολύ χαμηλές. Χρειάζεται να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για τα προγράμματα τα οποία βοηθούν τις ε, νέες γυναίκες και τους νέους όπως ε, το πρόγραμμα Youth on the Move. Για τις γυναικείες επιχειρήσεις και την αυτόνομη εργασία. Και γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε και η Επιτροπή μας πρέπει να δώσει σαφέστερες υποδείξεις. διαπιστώσαμε ότι δίνοντας κίνητρα στην σύσταση γυναικείων επιχειρήσεων, ε, κυρίως στον τομέα της κοινωνικής ε, ε, οικονομίας και στις no profit οργανώσεις, διαπιστώσαμε ότι εκεί δημιουργείται απασχόληση όταν βλέπουμε ότι οι δημόσιες θέσεις εργασίας κλπ δεν υπάρχουν. Επίσης, η Κομισιόν θα μπορούσε να διαπιστώσει πώς χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει μια τεράστια δυσκολία σε πολλές χώρες για την χρήση των, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και δεν χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκοί ε, πόροι διότι δεν υπάρχει η εθνική συγχρηματοδότηση. Δεν θα μπορούσε στον τομέα της ε, συγχρηματοδότησης να μειώσει αυτά τα ποσοστά η Ένωση τουλάχιστον σε μια αρχική φάση του σχεδίου για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά τα προγράμματα και δεδομένου ότι αυτά τα προγράμματα είναι περισσότερο περιφερειακά και όχι εθνικά. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος, κυρία Κώστα. Η κυρία Μπαλτσάνη έχει το λόγο και πάλι. Grazie per gli interventi. Mi sembra di cogliere da questo, da questo primo incontro. Ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις. Μου φάνηκε να διαπίστωσα έναν καμβά σε αυτή την Επίτροπη. Οι πέντε στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας συνδέονται στενά με την προβληματική των γυναικών και κυρίως την προβληματική της εργασίας. Η εργασία είναι κάτι το ευρύ πέρα από την απασχόληση, αφορά στη σύσταση επιχειρήσεων, στην ειδικευμένη εργασία. Αυτή η πρώτη προσπάθεια συμμετοχής στη διαδικασία του προϋπολογισμού απαιτεί να ορίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τις προτεραιότητες αυτής της μεγάλης στρατηγικής που είναι τόσο συνδεδεμένη με την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα θέμα που επανέρχεται ιδιαίτερα πιεστικά σε περίοδο κρίσης πρέπει να ε, ανακάμψουμε το ΑΕΠ και την απασχόληση. Και για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται συμμετοχή όχι μόνο στην οικονομική και κοινωνική ζωή αλλά και στον πολιτικό βίο. Διότι η έλλειψη συμμετοχή στον πολιτικό βίο έχει σοβαρές επιπτώσεις και στα οικονομικά. Αυτό είναι ένα σημαντικό ε, σκέλος της στρατηγικής 2020, κυρίως σε μια φάση κρίσης που θα πρέπει να μας οδηγήσει να ανακαλύψουμε ποιες είναι οι χαμένες μας ευκαιρίες. Βελτίωση των συνθήκων για τη συμμετοχή στο δημόσιο βίο. Όλα αυτά συνδέονται και με την διαχείριση του οικογενειακού βίου να διαμορφώσουμε τους όρους για να συμβεί κάτι τέτοιο. Χρειάζονται επενδύσεις φυσικά και των κρατών μελών για να αποσυρθούν τα εμπόδια. Αυτή η εργασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για αυτή μας την Επίτροπη και για τις προοπτικές 2020 που αφορούν κυρίως εμείς ε, άρουμε τεμπόδια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπαλτσάνη για τις πληροφορίες, για το γεγονός ότι ήρθατε εδώ να συμμετέχετε στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Σενκλέρ... Έχω ένα διαδικαστικό, κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε ότι προσπαθώ να δω τι θα κάνει την πράγμα και στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθώ να οργανώσω τη, τη, δουλειά μου. Ε, το πρόγραμμα που το έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το Ιράν θα συζητήσουμε στα, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι συνάδελφοι ε, επίση μπερδεύτηκαν. Ε, Μήπω θα πρέπει να χτενίσει το γνωδιάγμα να είναι πιο βολικό, πρόεδρος. Ναι, την υπόψη αυτό το οποίο είπατε και είναι αλήθεια ότι είναι σημαντικό να προσπαθούμε ε, να ε, τηρούμε το χρονοδιάγραμμα όπως το προβλέπει η Μέρση Διάταξη. Όμως ε, σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής δυστυχώς χρειάστηκε να ασχοληθούμε με μια αλλαγή. Μια αλλαγή στο πρόγραμμα που θα κάνουμε, την κυρία Λάγκμπακ. Είναι κάτι το οποίο το προβλέπαμε στη Μέση Διάταξη Όμω η κυρία Λάγκμπακ είχε κάποιο πρόβλημα με το αεροπλάνο και ε, αποφασίσαμε να αλλάξουμε την μέση διάταξη και γι' αυτό το λόγο είχαμε αυτή την αλλαγή. Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Σιγκλέρ. Αρχή-αρχή όταν άρχισε η συνεδρίαση το αποφασίσαμε. Πρόκειται για γεγονός εξαιρετικής φύσεως και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Då går vi alltså till... συνεχίζει. Άρα, πάμε τώρα στο σημείο αριθμούν 6 που αφορά το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Είναι θέμα το οποίο σχετίζεται και με αυτό που τώρα μόλις συζητήσαμε. Για διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ε, για το πόσο σημαντική είναι η δραστηριότητά τους για την εισοδό των φύλων η κυρία Οβίρ το έχει αναφέρει, δεν είναι εδώ, αλλά η κυρία Νικολά ε, θα μας ενημερώσει από πλευρά τη εισηγητρίας. Ναι, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς η συνάδελφός μου δεν είναι εδώ παρούσα και εγώ προσπαθώ να παρουσιάσω την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Οβίρ. Ελπίζω ότι οποιασδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις θα μπορέσει να τις διεξέλθει η κυρία Οβίρ όταν θα έρθει εδώ. Πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η κυρία Οβίρ προσπάθησε να έχει μία σειρά ορισμών που είναι πολύ σημαντικές για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τμήμα των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Περιλαμβάνουν επίσης και την, ε, τις υγειονομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες οικουμενικού χαρακτήρα. Είναι υπηρεσίες που δίδονται άμεσα στο ενδιαφέρομενο άτομο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην συνοχή και τη συμπερίληψη και όλα αυτά απαρτίζουν ένα σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα. <coughs> Τίθεται εδώ και το κεντρικό θέμα της σχέσης μεταξύ του οικονομικού και του κοινωνικού τομέα. Που για μας είναι και το ουσιαστικότερο θέμα στις τωρινές συνθήκες, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εξισορρόπηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως σε εποχής οικονομικής κρίσης και λιτότητος προϋπολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ καλούς ορισμούς για τα θέματα αυτά η Κομισιόν το προηγούμενο Οκτώβριο αναφερόμενη στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος είπε ότι δεν πρόκειται να υποβάλει νέες προτάσεις στα θέματα αυτά. Ο κύριος Ντερόσα πρότεινε να υπάρξουν δομές οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος να αντιμετωπιστούν χωριστά στους κανόνες δημοσίων προμηθειών. Και ανέφερε επίσης ο κύριος ε, Τερόσα ότι πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση και των κανόνων σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή εμπλεκομένων. Η γνωμοδότηση της κυρίας Σόβιρ τονίζει και να ληφθούν υπόψη περισσότερο τα θέματα αυτά από τις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ότι οι περικοπές από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μην βλάψουν την οικουμενικότητα της προσβασιμότητας της υπηρεσίας αυτές δύο και θα πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει μια οικονομική συνεισφορά του κράτους όπως και την εποχή των παχαιών, των παχαιών αγελάδων. Τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβουν το λεγόμενο gender budgeting, την κατανομή του προπολογισμού αναφύλω σε όλες τις πολιτικές τους. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 22 Μαρτίου και η Επιτροπή μας θα ψηφίσει στις 20 Απριλίου και φυσικά περιμένω να το επιβεβαιώσετε αυτό κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ τα μάλα. Προσπάθησα να κάνω ό,τι το ανθρωπίνο δυνατό εξονόματος της Κυρία Σοβίρ και όταν έρθει η κυρία Οβίρ ελπίζω τα ερωτήματά σας θα έχουν μια πλήρη απάντηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Η κυρία Σελεύσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι σήμερα στην Επιτροπή μας έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Αυτέ είναι οι υπηρεσίε οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως από άτομα τα οποία βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, από άτομα τα οποία έχουν πληγεί και από την οικονομική κρίση. Όταν μιλάμε για κοινωνικές υπηρεσίες, μιλάμε για σπίτια, για στέγαση, για σπίτια για τους ηλικιωμένου, τους ανάπηρους, για τις γυναίκες που είναι θύματα βίας, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αλλά και κέντρα ε, υγειονομικά, καπή και άλλους φορείς που παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες. Όχι με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά ακολουθώντα τις τοπικές παραδόσεις, την ανάγκη αλληλεγγύης και την ανάγκη φροντίδας των ασθενεστέρων. Ένα χαρακτηριστικό αυτών των <clears throat> υπηρεσιών είναι ο γενικός και οικουμενικός τους χαρακτήρας και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των μεμονωμένων ατόμων. Ο ρόλος αυτών των υπηρεσιών είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι μέσω αυτών αντιμετωπίζουμε τον αγώνα κατά της διακρίσεως, την ισότητα των φύλων, είναι ένα στοιχείο υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, βοηθούν την κοινωνική συνοχή, ανεξάρτητα από τον πλούτο των πολιτών και υποστηρίζουν και την ανθρώπινη υγεία. Συζητούμε τον τελευταίο καιρό πώς θα πρέπει να καθορίσουμε τις υπηρεσίες αυτές ως οι οικονομικές υπηρεσίες ή όχι. Και επίσης για το αν θα πρέπει να υπόκεινται στην νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στον στόχο αυτών των υπηρεσιών και να τονίσουμε το ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και στους κανόνες ανταγωνισμού και ποιε υποστηρίζουν την οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή και επομένω θα πρέπει να είναι εκτό του πεδίου εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία. Για να αντιμετωπίσω τώρα ε, άμεσα την γνωμοδότηση τη κυρία Οβίρ εγώ υποστήριζω αυτά που λέει ότι οι υπηρεσίε για τη φροντίδα των παιδιών πρέπει να γίνουν πάρα πολύ πιο προσβάσιμε και πιο ε, φτηνέ. Έχουμε κάνει λοιπόν πολλέ προσπάθειε προ την κατεύθυνση αυτή και είναι η θαυμάσια ευκαιρία αυτή η έκθεση για να τονίσουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Δεν πιστεύω όμω ότι αυτή η έκθεση είναι θεματικά επαρκή για να συζητηθεί η ψαλίδα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πολλαπλά τέτοια φαινόμενα τα έχετε δει αγαπητές συνάδελφοι και τα έχετε αναφέρει στην Ολομέλεια σε άλλες ευκαιρίες. Η συγκεκριμένη αυτή δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να θίξουμε τέτοιου είδους συζητήματα. Στην Πολωνία, στον κοινωνικό τομέα, 90% των εργαζομένων είναι γυναίκες και 10% άνδρες. Ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και την χρηματοδότηση των κοινωνικών υποθέσεων στο επίπεδο πριν από την κρίση και αυτό είναι το κέριο στοιχείο του εγγράφου. Αν υπάρξει μείωση της χρηματοδότησης, οι γυναίκες θα γίνουν διπλά θύματα γιατί θα υπάρχουν λιγότερες πηγές χρηματοδότησης για την φροντίδα των παιδιών και έτσι οι γυναίκες δεν θα μπορούν να δουλεύουν. Ο τομέα των υπηρεσιών επίση δημιουργεί πολλή εργασία για τι γυναίκε, όπω ανέφερε και η κυρία Οβίρ στο σημείο 5. Δυστυχώ λοιπόν δεν είναι παρούσα η κυρία Οβίρ. Θα ήθελα το ερώτημα αυτό να το διαβιβάσετε. Και έχω ένα πρόβλημα με το σημείο 2 της γνωμοδότησης με την ε, έκφραση ενεργητικές στρατηγικές για την ευμάρεια. Θα ήθελα η κυρία Οβίρ να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η φράση γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω και θα ήθελα και η γραμματεία να λάβει υπόψη το γεγονός ότι στη μετάφραση προς τα πολωνικά υπάρχει μια, ένα σφάλμα. Μετά από τις λέξεις για το μέλλον των υπηρεσιών δεν υπάρχει λέξη κοινωνικός. <clears throat> Υπάρχουν απλώς υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος αλλά δεν έχουν τη λέξη κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος, η κυρία Μπάστου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Προσπαθήσω να είμαι ως να τον πιο σύντομη, γιατί το θέμα αυτό των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολλές φορές. Θέλω να σας πω ότι στη γνωμοδότηση αυτή είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή διάκριση σε σχέση με τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος αφενός και τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Γιατί ο στόχος μας στην Επιτροπή μας είναι να συμβάλλουμε ώστε με μεγάλη σαφήνεια η έκθεση του κυρίου Τεχώσα να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει με σαφήνεια τι είναι ακριβώς οι κοινωνικές υπηρεσίες μέσα στον τομέα γενικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, δηλαδή ποιες είναι αυτές οι οποίε άπτονται πιο άμεσα των αναγκών του πληθυσμού και παίζουν ένα μεγαλύτερο ρόλο στην εξασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνενοχής στις κοινωνιτές μας. Κάθε χώρα, κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του νομοθεσία για τα θέματα αυτά για να αντιμετωπίσει και να νομοθετήσει σε σχέση με τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Αυτό το οποίο μας απασχολεί εμάς είναι σε αυτές τις στιγμές οικονομικής κρίσης και πρέπει να από την εκθεσή μας να μην υπάρξει περιορισμό στην πρόσβαση και ιδίως στην ποιότητα και στο τίμημα για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, οι οποίες καλύπτουν και τις βασικές ανάγκες των πληθυσμών μας. Από την άποψη αυτή, εγώ θέλω να υποστηρίξω τις ε, παρατηρήσεις της προλαλήσας σας, συναδέλφου, που τονίζει ότι θα πρέπει κάποιες από τις ε, παρατηρήσεις που αναφέρονται στη γνωμοδότηση της κυρίας Σοβίρ να αντιμετωπιστούν και αυτές μέσα στην έκθεση αυτή. Παραδείγματος χάρη το θέμα της ανισότητος των αποδοχών. Στα θέματα της ε, παιδείας, της ε, υγειονομικής περίθαλψης, της πρόσβασης στο καθαρό νερό κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να περιληφθούν στην έκθεσή μας για να αντιμετωπίσει σωστά όλα αυτά τα ζητήματα σε μια εποχή κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Θέλει η κυρία Νικολάη να πει κάτι για όλα αυτά. Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση στα ερωτήματα των συναδέλφων μου για το σημείο 2. Μπορώ όμως να κάνω κάποιο μικρό σχόλιο για την ε, διάκριση μεταξύ κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών. Εγώ συμφωνώ πλήρως με την ε, κυρία Μπαστός, η οποία τόνισε ότι υπάρχουν δύο ειδών υπηρεσίες. Έχει να κάνει με τις γενικές κατηγορίες και τις ειδικέ κατηγορίες, αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις κοινωνικές υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντος. Και σύμφωνα απόλυτα για αυτό το θέμα με την προλαβή σα. Για, το, για την ανισότητα αμοιβών στις κοινωνικές υπηρεσίες και την υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των δύο φύλων. Δεν ξέρω αν αυτή η έκθεση είναι ο πιο πρόσφορος τόπος να αναφερθούμε στο θέμα αυτό, αλλά αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί βλέπουμε στα κράτη-μέλη να υπάρχει μια θηλυκοποίηση ορισμένων επαγγελμάτων. Τα θέματα της υγειονομικής περίθαλψης, παραδείγματος χάρη. 70% των εργαζομένων στον τομέα αυτό είναι γυναίκες. Και δυστυχώς στα κράτη-μέλη οι αμοιβέ στον τομέα αυτό, τον κοινωνικό και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι ελκυστικά δεν είναι ελκυστικέ οι αποδοχές αυτές και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε γιατί για αυτού του είδους τι υπηρεσίες η μόνιμη παρουσία και η απόδοση αυτών που εργάζονται στον τομέα αυτό είναι κεφαλαιόδους σημασία. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο να αναφερθούμε στην ψαλίδα αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα υπόλοιπα ερωτήματα νομίζω θα δώσει μια απάντηση η κυρία Οβίρ στην επόμενη συζήτηση που θα έχετε επί τη βάση του εγγραφού εργασίας. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. information om tidtabellen. τώρα, κάποια ενημερωτικά. 22 Μαρτίου το μεσημέρι εκπνέει προθεσμία της τοπολογίας και θα ψηφίσουμε στι 20 Απριλίου και στην Επιτροπή Απασχόληση το Μάιο. Ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η ψήφιση στην Ολομέλεια. Mm. Συνεχίζουμε τη μέση διάταξη και πάμε στο σημείο υπαρθμών 7. Η πέμπτη έκθεση Επιτροπή για τη Συνοχή και η πολιτική συνοχή μετά το 2013. για την ε, Επιτροπή μας, η συντάκτης ο κύριος Σιμάνσκι και στον οποίο θα του δώσω το λόγο. Πέστε μας δύο λόγια. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω τα εξής στοιχεία της εξής προτάσεις. Έχετε λάβει το έγγραφο, αλλά μπορώ να σας ε, προσθέσω τις δικές μου παρατηρήσεις. Νομίζω ότι η πέμπτη έκθεση για την Επιτροπή Συνοχής πάρα πολύ λίγο συζητά τα θέματα ισότητας των φύλων, αλλά και ίσων ευκαιριών. Επομένως, εδώ διδέχεται μεγάλη βελτίωση αυτό το κείμενο και εμείς επομένως να υποβάλουμε κάποιες προτάσεις για τροποποίηση του κειμένου και έτσι να φυγεί περισσότερο το θέμα της ισότητας. Αλλά το θέμα της συνοχής του 2013 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη περισσότερο. Είναι θέμα ισότητας των φίλων. Έχω συγκεκριμένε προτάσει στο σχέδιο κειμένου που σα έχω βάλει. Ασχολούμαι συγκεκριμένα με τα εξή. Αυξημένη οικονομική υποστήριξη, πληκοδότηση κάποιων δράσεων, τόσο ώστε γυναίκε και οι άντρε να μπορέσουν να συνδυάσουν οικογενειακό βίο και επαγγελματικό βίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει αποτυπωθεί από τα όσα συζητήσαμε πριν. Ιδίω όσον αφορά τι υποχρεώσει των γυναικών για δουλειά και για το σπίτι. Και είναι και θέμα επίση κοινωνική ασφάλιση. Τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί σε μια σειρά χωρών μελών ε, ε, υπάρχουν διαφορετικέ λύσει. τι θα κάνει η Ευρώπη, γιατί μια γυναίκα πολλέ φορέ υποχρεώνεται, αναγκάζεται να θυσιάσει την οικογενειακή ζωή, όμως ε, δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να επιβιώσει εάν κάτι το συμβεί. Επίσης, αυτό μας παραπέμπει και στο πρόβλημα της φτώχειας για τις γυναίκες. Επίσης, ε, έχουμε το θέμα της επαγγελματικής ε, δραστηριότητας και την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εδώ έχω μια σειρά προτάσεων. Ας πούμε, μιλώ για συγχρηματοδότηση και κάποιε πρωτοβουλίες που αφορούν τις γυναίκες των 45. Προγράμματα ισοβίας κατάρτισης, μια που η παιδεία εδώ είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να επενδύσουμε σε προγράμματα κατάρτιση, σε επαγγελματικού προσανατολισμού και για τι γυναίκε που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα παρακαλώ να λάβετε υπόψη αυτή την πρόταση, την ισόβια κατάρτιση εννοώ. Επίσης, θα ήθελα να έχω μια τροπολογία. Μια τροπολογία στον που δουλεύουν σε συνθήκες ε, ιδιαίτερα ευάλωτες. Πάρα πολλοί δεν μπορούν να δουλέψουν σε πλήρη απασχόληση, γιατί εδώ πέρα είναι το θέμα κάποιων προτύπων, κάποιων συνθήκων υπό τι οποίε ε, δουλεύουν κάποιε γυναίκε και τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ σταθερά. Σε πάρα πολλέ χώρε οι γυναίκε αναγκάζονται να δουλέψουν σε κάποιο ελευθερίο επάγγελμα. Δηλαδή, παρετούνται από την δουλειά που είχαν προηγουμένω και κάνουν τώρα την ίδια δουλειά σαν ελεύθεροι επαγγελματίε. Αυτό με εξοικονομεί δαπάνε, αλλά επιδεινώνει το βιωτικό του επίπεδο. Πρέπει αυτέ οι νίκε να πληρώνουν τι ε, εισφορέ του και επίση όταν αυτές οι γυναίκες γίνουν μητέρες, υφίστανται αυτή την υποβάθμιση. Εδώ θέλουμε να προάγουμε τις άριστες πρακτικές και όχι απλώς να νομοθετούμε. Επίσης, να μελετήσουμε το τι θα γίνει στο μέλλον σε αυτή την πολιτική της συνοχής, πώς θα βοηθήσει για σταθερές ε, εργασίες, αποκεντρωμένες διαδικασίες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ξέρουμε ότι ο ολλανδοί Πασοτική είναι και μπαίνουν σε αγορά εργασίας. Και όλα και περισσότερες είναι οι φτωχέ γυναίκες, αυτέ που μαστίζονται τη φτώχεια και πάρα πολλέ βρίσκονται κάτω από το κατόφλι της ανέχειας. Άρα Ήδη έχουμε συζητήσει τα θέματα της μελών διακρίσεων, κάτι το οποίο αφορά κυρίω τον περιοδο 2000-2006. Άρα δεν αποτυπώνεται εδώ η κατάσταση στα νέα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και όσον αφορά την πολιτική τη συνοχή, οι εμπειρίε πολλών κρατών μελών θα πρέπει να αναλύονται. Ιδίω λαμβάνοντα υπόψη το τι γίνεται στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Παρακαλώ, ε, όποιο θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο μου και να μου μας πει την, ε, τι, τι, τι, έχει να προτείνει. Και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τροπολογία μας και νομίζω θα βελτιωθεί έτσι η κατάσταση των γυναικών. Ευχαριστώ για αυτές τις ε, πληροφορίες και για τις διάφορες προτάσεις πριν ε, έκθεση είναι θέματα πολύ σημαντικά τα θέματα της ε, <coughs> πολιτικής συνοχής ε, για τις γυναίκες, για την απασχόληση. Τώρα έχουν το λόγο οι συνάδελφοι της Επιτροπής. Αν δεν θέλει κανείς το λόγο, όπως είπε και ο κύριος Σιμάνσκι, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί του και να παρουσιάσετε τις ε, το, παρατηρήσεις σας για να βελτιώσει το κείμενό του. 22 Μαρτίου στις 12 λίγη προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Η ψηφοφορία 20 Απριλίου και η Ρέτζη θα ψηφίσει από 9 ως 12 Μαΐου για να περάσει στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Σιμάνσκι και πάμε στο επόμενο σημείο. Μεγάλη μου ευχαρίστηση που υποδέχομαι την κυρία Λαγκμπακ που θα μας μιλήσει για τις εργασίες και το, προς, το επόμενο πρόγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να έχουμε τις ε, πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας του 2011 και να ενημερωθούμε για το ποιες είναι οι παρούσες εργασίες του Ινστιτούτου. Ε, ευχαριστούμε την κυρία Λάντμπακ και της δίνουμε ευθύς αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσω τη δουλειά μας και και βεβαίω είναι για την πρώτη φορά που επιτέλους θα φανεί η δουλειά μας. Πριν από λίγες εβδομάδες προσπαθούσαμε εμείς να εκπονήσουμε κάποια δείγματα, κάποια, να προσφέρουμε τις ενδείξεις της ε, κατάστασης για τις ε, ανισότητες. Και κατάσταση είναι τέτοια που έχουμε 2% υπουργού ε, γυναίκες και 98 άντρες 5% ε, 10% διπλωμάτισες το έχουν αρχίσει και οι άντρε να παίρνουν γονική άδεια και έχει αλλάξει κατάσταση. Όμω η διαφορά είναι το ότι τώρα ξέρουμε το τι συμβαίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε και μπορούμε να πάρουμε συγκεκριμένε πληροφορίε. Δεν ξέρω τι γίνεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, πώς ε, διαδίδονται οι άριστες πρακτικές. Και γι' αυτό και συγκροτήθηκε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο μας από εσά. Θέλουμε να σας ε, ευχαριστήσουμε και σύντομα μπορεί να σας παρουσιάσω το τι έχουμε επιτελέσει. Αργήσαμε να σας ε, στείλουμε το υλικό αυτό, δυστυχώς. Να σας πω τι έγινε για το 2011 πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει εγκριθεί. Και εκπονούμε τώρα το πρόγραμμα για το 2012. Σε επαφή με την Κομισιόν, με το Διοικητικό Συμβούλιο, για να δοθεί έγκριση πριν δημοσιοποιηθεί. Έχουμε επομένω αυτό το κέντρο αριστεία για την ισότητα των φύλων. Και έτσι προχωράμε, προσπαθώντας να εκπονήσουμε έναν ορισμό. Δηλαδή να, να περιχαρακώσουμε το σκοπό του Ιδρύματος. Πριν από έναν χρόνο εγκατασταθήκαμε στο Βίλνιους τον Δεκέμβριο και είχαμε τον κύριο Σπίτλερ και άλλους ε, που μας βοήθησαν στα εγγένεια μετά τον Ιούνιο λίγο μετά από έξι μήνες αποκτήσαμε διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία όπως και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Πρώτος του Κοινοβουλίου επίσης για και τα εγγένεια. Είδα ότι αποκτήσαμε και λογότυπο. και έδωσε η Επίτροπος Ρέντινγκ κάποια βραβεία, όπως κάποιοι, κάποιοι δάσκαλοι από την Γαλλία και κάποιοι από την Πολωνία, λάβανε το δεύτερο βραβείο. Επίσης οργανώσαμε ένα σεμινάριο εκεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τη στρατηγική της για την ισότητα των φίλων. Και ε, ε, καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες. Δεν μπορέσουμε να έχουμε τελικά ένα για το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όποιον χρειάζεται ως ίδρυμα. Πολύ σημαντικό και αυτό για τη δουλειά μας. Επίσης, δημοσιεύσαμε ένα καλαντάριο δραστηριοτήτων και πρόκειτο για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σταρ, και αυτό, από τις Μαλτές και τις Εφημερίδες. Ήδη πετύχαμε να υλοποιηθεί κάποιο σχήμα συνεργασίας όσον αφορά τις αδελφές υπηρεσίες. Δηλαδή, να δούμε πώς υπάρχει συνέργεια και όχι επικάλυψη. Άρα έχουμε τρεις άλλες συγγραφείς υπηρεσίες με τις οποίες εργαζόμαστε. Να γίνει πραγματικότητα η ισότητα θέλουμε. Για όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι το όραμά μας. Εμείς προχωρούμε στην επιτυχία του στόχου, μην ξεχνώντας πόσο σημαντικό είναι αυτό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να υλοποιηθεί αυτός μας ο στόχος. Ελπίζω δεν θα πάρει άλλον έναν αιώνα, όπως περιμέναμε έναν αιώνα για τις κατακτήσεις αυτές. Ε, εντάχει να σας πω το ότι μετά το 2010 έχουμε τις προτάσεις μας όσον αφορά το από πού θα προέρχονται οι υπαλληλοί μας. Επίσης να δείτε με τι ρυθμούς αυξήθηκε η δουλειά μας μετά το δεύτερο εξάμεινο πέρσι. Αυξήθηκε το προσωπικό, τις έχουμε όλους όσους χρειαζόμαστε σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταδείξει το 2010. Κάτι άλλο το οποίο θα σας δείξει πώς λειτουργούν τα προγράμματα που έχουμε για τη δουλειά μας. Γιατί έχουμε, είπαμε, προσωπικό από παντού, ασχολούνται με μελέτες και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε απορροφήσει το 60% του προϋπολογισμού μας. Θα είναι τα πράγματα πιο εύκολα το 2010 από το 2010. Επίσης, εδώ σας έχουμε και ένα γράφημα σε σχέση με το ε, τι κάνουμε, πώς σχεδιάζουμε τη δουλειά μας. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό κέντρο αριστείας εδώ. Οπότε έτσι <coughs> θα αναλύεται και θα διαδίδεται η δράση μας στους βασικούς εμπλεκομένους. Τα τρία θεσμικά οργάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και επίση επί το παρόντος, το πρόγραμμα εργασίας έχουμε τους δείκτες του Πεκίνου. Υποπτία, ανθιώρηση και έχουμε αυτό τον δείκτη ισότητας των φύλων. Γίνεται δηλαδή των καλών πρακτικών. Και τα βασικότερα θέματα που αφορούν τα δύο φύλλα, αυτή η διαδικασία επομένω. Μαζεύουμε στοιχεία. Στατιστικά για διάφορε πρακτικέ, ό,τι στοιχεία χρειάζονται, τόσο ώστε αυτά όλα να τα έχει το κέντρο έρευνα. Οπότε μέχρι το τέλο του 2011 θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε κάποιε από αυτέ τι πληροφορίε για να μπορέσουμε να προβούμε σε κάποιε δημοσιεύσει όμως με ανάγκες. Ακόμα είμαστε στη φάση της περισυλλογής, αλλά αλλού πούμε πιο γρήγορα, αλλού πιο αργά. Για κοιτάξτε τώρα το πρόγραμμα του 2011, πρόγραμμα εργασία, έχουμε εδώ κάποια συγκρίσιμα υγεία αξιόπιστα. Αυτή είναι η βασική δείκτες μας οδηγούν στο να δούμε τι συνδεδομένα θα συλλέξουμε, να γίνει κάποια αναθεώρηση και να προχωρήσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου. Επίσης και με κάποια πιλωτικά προγράμματα ασχοληθήκαμε. Ακόμα και αν το θέμα της βίας των γυναικών δεν προκρίθηκε από τα κράτη-μέλη Και είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε Τι ενδιαφέρει τα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανθρώπινα δικαιώματα, γυναίκε, ΜΜΕ, ακόμα δεν έχουμε ασχοληθεί, γιατί πρόκειται για ε, ένα ε, νέο τομέα, έχουμε προετοιμάσει αυτέ τι ε, μελέτε που θα μα απασχοληθούν στο εγγύς μέλλον. Πολωνέζικη, Δανέζικη Κυπριακή Προεδρία στην Τρόικα. Σύνομα θα έχουμε τα αποτέλεσμα και αυτή τη μελέτη όσον αφορά την συμφιλίωση. Είναι κάτι το οποίο ασχολείται κυρίως η Πολωνική Προεδρία. Γυναίκες και περιβάλλον. Και αυτό είναι άλλο θέμα, δεν έχουμε τους σχετικούς δείκτες και θα, εδώ θα είναι πάρα πολύ σημαντικό πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε τελικά πού θα καταλήξει η έρευνα. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσει κανείς όχι μόνο θεσμικά οργάνωση, αλλά όλοι οι χρήστες με αυτά τα δεδομένα, τα στατιστικά, να πιστεύουν ποια είναι τα προβλήματα. Όπως σας είπα, η γυναίκα και η οικονομία, η γυναίκα και το περιβάλλον. Είναι οι δύο μέρες που σας είπα έχουν ξεκινήσει, συμπληρωματικές, και θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση μιας έκθεσης της Προεδρίας. <coughs> Για το 2012 τώρα. Μου προγραμματίσει να στοιχήσουμε την ε, αρρωγή προς την Προεδρία. Δεν ξέρουμε τι έχει διαλέξει η Κύπρος και τι η Προεδρία, αλλά είπαμε σε όλη διαλέξη η Προεδρία να περισυλλέξουμε δεδομένα και έτσι να βοηθήσουμε στην σύνταξη κάποιων συμπερισμάτων τώρα. Έχουμε το δίκτυο της ισότητας των φύλων και τελικά να έχουμε κοινά κριτήρια για να μπορεί κανείς να δει αν υπάρχουν ανισότητες αδικίες στα Πέρσι έγινε μια τέτοια μελέτη. Τι κατάφερε κάθε κράτος μέλος. Τι ισχύει το στα μέλη για αυτό το δίκτυο. Υπάρχουν όμως πολλοί δείκτες από τον ΩΣΑ, από, από άλλους οργανισμούς, τον ΟΗΕ, οπότε θα πρέπει να συγκρίνουμε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για να δούμε τι θα προτείνουμε. Με αυτό που αποφάσισαν για την έννοια του δίκτου Τα κρατημέλη, οπότε τώρα ολοκληρώνεται αυτή η μελέτη, η πρώτη μελέτη. Να έχουμε κάποια κάποιους ε, ε, ε, για να δούμε την αξιοπιστία των δεδομένων και για τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται την αρχική πρόταση. Και υπάρχουν κάποιες επίσης οι οποίες συνδέονται με τη στρατηγική της Κομισιόν για να μπορέσουμε να διακριβώσουμε σε ποιο βαθμό αυτοί οι δείκτες είναι επαρκείς για τη μέτρηση της πρόοδου σε αυτές τις περιπτώσει και σε αυτές τις περιοχές. Επίσης προσπαθούμε να δούμε πώς ε, λειτουργεί μεταλαμπάδευση των πρακτικών στον τομέα αυτό και το, η, το mainstreaming και τα θέματα του φύλου είναι ένας κεντρικός τομέας. Έχουμε πολλές ιδέες για τα θέματα αυτά. Για το ποιε θα μπορούσαν να είναι οι πιλωτικές περιοχές και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Αλλά το θέμα του mainstreaming είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές παραμελείται και παραγνωρίζεται και παραπετάται και δεν τη χάνει τη πρέπουσα προσοχή. Και επομένω θέλουμε να απτύξουμε περισσότερε ικανότητε για το τομέα αυτό. Και από πέρσι έχουμε συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία με τη μελέτη η οποία έγινε για τις υπάρχουσες πρακτικές και αυτή θα είναι βέβαια από τις πρώτες μελέτες που θα παρουσιαστούν μέχρι το τέλος του 2011. Έχουμε όμως και τις ε, βέλτιστες πρακτικές. με κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους φορείς σε όλη την Ευρώπη. Γιατί διαφορετικά κράτη-μέλη έχουν διαφορετικέ ενδιαφέρουσε προσεγγίσει και άμα δεν τι ξέρετε, δεν μπορείτε να τι μετρήσετε, δεν μπορείτε να τι χρησιμοποιήσετε, δεν μπορείτε ούτε να τι παραγνωρίσετε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα για μας λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλουμε επίση να περιλάβουμε ω παράδειγμα βελτίστων προκτικών, πρακτικών είναι και η μελέτη κατάρτιση στοιχείων για τους φορείς που ασχολούνται με τα θέματα του φύλου μέσα στα πλαίσια της εργασίας μας θέλουμε να έχουμε και μια ομάδα αναφοράς ανδρών για να δούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται η προοπτική του φίλου και πώς εισάγεται στα διάφορα θα Προσπαθούμε τώρα να προσκαλέσουμε τις οργανώσεις ανδρών στην Ευρώπη να συμμετάσχουν στην εργασία του δικτύου μας γιατί θα έχουμε και ένα ανδρικό δίκτυο. Ένα δίκτυο ένα δίκτυο για τους άνδρες που εργάζονται για την ισότητα των φύλων. Θέλουμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η προσέγγισή τους. Θα δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν το Ινστιτούτο μας νομίζω θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει για να καταδείξει ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Κάναμε και μία επίσης μελέτη για τα στερεότυπα και τις αφηγηματικές πρακτικές πώς μέσα σε μια οικογένεια, πόσα μέσα στη βάση, η αντίληψη του φίλου σε αφηγηματικό επίπεδο αποτελεί παράγοντα προσδιορισμού της επερχόμενης πολιτιστικής αντιμετώπισης των γενεών που ακολουθούν και θέλουμε να συνδέσουμε λοιπόν τα στερεότυπα και την επιλογή επαγγέλματος τις καριέρες που επιλέγουν οι νέοι, τα σουσούμια τους και τα χούγια τους. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και να τα απεικονίσουμε. Για τα μελλοντικά σχέδιά μας έχουμε επίσης κάποιες προτάσεις για το 2012. Σκεφτόμασταν εργαλεία mainstream και βέλτιστες πρακτικές να θεωρήσουμε ότι η εκπαίδευση για τα θέματα του φύλου είναι ένας τομέας όπου είναι φανερό ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ακόμα να προχωρήσουμε και από το ευρωπαϊκό επίπεδο προς το <clears throat> τοπικό επίπεδο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συλλέξουμε δεδομένα για αυτούς οι οποίοι εκπαιδεύουν για τα θέματα του φύλου, να υπάρχει μια βάση δεδομένων ε, επιγραμμική στο διαδίκτυο για να μπορούμε να γνωρίζουμε όλα αυτά τα οποία πράττουν αυτοί οι εκπαιδευτές και θέλουμε επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές και θέλουμε εμείς να διοργανώσουμε και ένα σεμινάριο, μια συνδιάσκεψη, όπου θα εξετάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης σε σχέση με το φύλλο που θα παρουσιαστούν σε μια κοινή διασκέψη, όχι μόνο με τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό, αλλά και σε σχέση με αυτούς οι οποίοι θα ενδιαφερόντουσαν να τύχουν τέτοια εκπαίδευση και φυσικά εκεί θα εξετάσουμε και τα θέματα της ποιότητα και το επίπεδο ποιότητα. Αυτό το οποίο επίσης θέλουμε να κάνουμε επί τη βάση <clears throat> του έργου μας το 2011 είναι να συλλέξουμε και στοιχεία βελτίστων πρακτικών στον τομέα της συμφιλίωσης γιατί αυτό είναι σημαντικό και σε σχέση με τη θέση των γυναικών στα θέματα της οικονομίας και για την βία που στηρίζεται στη διάσταση του φύλου. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτά τη στιγμή. Θα κάνουμε και άλλες μελέτες επίσης για να μπορέσουμε να περατώσουμε την εξέταση ορισμένων περιοχών που δεν έχουν ακόμα συνδεθεί μέθοδα, μέθοδοι και εργαλεία για την πρόληψη της βίας επί τη βάση του φύλου. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο προφίλ για το πώς μπορεί να βοηθήσει η μεταλαμβάνευση βελτίστων πρακτικών και η καλή εκπαίδευση. Επίσης, σε επίπεδο προϊόντων θέλουμε να έχουμε κάποιες δημοσίευσεις οι οποίες θα είναι <coughs> διαθέσιμες σε έντυπη μορφή και σε διαδικτυακή μορφή ώστε να μπορούν να τις αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται και να υπάρχουν και διάφοροι κατάλογοι ελέγχου για το πρακτέο τους τομείς αυτούς. Το 2012 επίσης <coughs> θέλουμε να περατώσουμε και τη διαδικασία δημιουργίας των δικτύων μας σε Ευρώπη για την διάσταση του φίλου να υποστηρίξουμε λοιπόν δίκτυα σε όλους του τομείς, αλλά όλους του θεσμούς, όλα τα άτομα τα οποία εργάζονται στον τομέα αυτό και θέλουμε να έχουμε και ένα ιδιαίτερο υποδίκτυο για την εκπαίδευση στα θέματα φύλου, ώστε να μπορούν να υπάρχουν ανταλλαγέ απόψεων και να μπορεί κανείς να προσθέσει πληροφορίε στα κέντρα ικανότητων, στα κέντρα πόρων για τη βία επιβάση του φύλου, για την φιλία και τον οίκο για όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν ώστε να μπορούν και οι άνδρες να συμμετέχουν στην ε, ε, αντιμετώπιση αυτών των ε, στοιχείων ώστε να αλλάξουν επιτέλους και την στερεοτυπική τους προσέγγιση. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο όπως είδατε στο πρώτο τμήμα. Αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε να έχουμε μικρές βιβλιοθήκες που να περιλαμβάνουν βασικά έγγραφα πολλές φορές είναι στοιχεία βιβλιογραφίας που δεν μπορούν να βρεθούν ούτε σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και επίσης η βιβλιοθήκη μας θα είναι κυρίως στο διαδίκτυο. Θα έχουμε συνδέσεις σε βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ώστε να μην επικαλυπτόμεθα μαζί τους αλλά όποιο έρχεται στο διαδικτυό μα θα βρίσκει αμέσω τη σύνδεση ώστε να μην χρειάζεται να ψάχνει στο διαβόλου τη μάνα και θα έχει τη δυνατότητα να έχει αμέσω πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την διάσταση του φύλου. Κέντρα γνώσης, αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο μα. Όλα τα εργαλεία, όλες οι μέθοδοι που αναπτύσσουμε, όλες οι εστιακές περιοχές και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων θα είναι ο χώρος όπου θα συνενώνονται όλα αυτά, θα συνενώνονται όλα τα υποδίκτυα θεσμικού χαρακτήρα, θα ανταλλάσσονται πληροφορίες και θα συνενώνονται οι βέλτιστες πρακτικές από τα διάφορα κέντρα ικανότητας. Τελευταίο στοιχείο. Μία μεγαλύτερη επίγνωση και καλύτερη επικοινωνία σε σχέση με τα θέματα του φύλου. Αυτό το οποίο θέλουμε να περατώσουμε είναι οι προσπάθειές μας να έχουμε καλύτερη στρατηγική σε εξωτερικό και εσωτερικό επίπεδο, εξωτερική επικοινωνία για την ισότητα των φύλων που άλλες φορές είναι συγκεκριμένο, άλλες φορές αφηρημένο θέμα και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το ερμηνεύει ο καθένα. Θα πρέπει να υπάρχει όμως σαφέ μήνυμα για κάθε ομάδα στόχου και έτσι η στρατηγική μας επικοινωνίας θα περατωθεί, θα οριστικοποιηθεί πολύ σύντομα, ώστε να μπορούμε να λέμε όλα αυτά τα στοιχεία, να είναι κατανοήσιμα και τα πραγματικά στοιχεία, αλλά και τα επιχειρήματα και τα εργαλεία και οι βέλτιστες προσπάθειες και όλα αυτά πρέπει να κάνει κάθε χώρα για να κλείσει το χάσμα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο επίσης ασχολείται με την επικοινωνία. Ξεκινήσαμε ήδη με τις γυναίκες της Ευρώπης πέρσι. Τώρα θα έχουμε μια ομάδα πόρων για τους άνδρες της Ευρώπης, για αυτούς που αξίζει να τους υμνεί και να τους επενεί κανείς. Αυτούς που έχουν παίξει ένα προεξάρχοντα ρόλο στην καριέρα τους, στη ζωή τους σε σχέση με την ισότητα των φίλων. Και έτσι θα προχωρήσουμε στη συνεργασία με τους εμπλεκομένους. Αυτά λοιπόν για τη συνέχεια. Όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία στο δίκτυο επικοινωνίας και τα σχέδιά μας είναι <clears throat> για το 2012 να έχουμε και άνδρες που θα βρουν τον τρόπο να παρουσιάσουν τους άνδρες, τους άνδρες οι οποίοι έχουν προσεγγίσει τις γυναίκες της Ευρώπης που έχουν παίξει ένα σημαντικό, ρόλο στην ισότητα των φίλων. Έχουμε ξεκινήσει ένα ηλεκτρονικό δελτίο και επίσης μια μορφή παρακολούθησης της ε, ισότητος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά θα συνεργαστούμε και με τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε περισσότερη συνεργασία, αλλά κυρίως με τους πιο εμπλεκόμενους στην Ευρώπη θα συνεργαστούμε. Και είναι ειλικρινής η ελπίδα μου ότι αυτά τα γελαστά άτομα τα οποία <clears throat> ήταν παρόντες στην έναρξη των εκδηλώσεών μας θα μπορέσουν κάποιοι από αυτούς να γίνουν και υπουργοί σε μερικά χρόνια και όχι απλώς να παρακαλούν τους υπουργούς για να βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Λάγκμπακ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Το λόγο τώρα οι συνάδελφοι της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κυρία Λάγκμπακ. Πολύ Χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα. Μίλησαμε προηγουμένως για την ανάγκη του να υπάρξει κάποια μορφή τακτικής ανταλλαγής απόψεων μαζί σας. Όχι και μόνο σε σχέση με την έγκριση του προϋπολογισμού ή για άλλα συναφή θέματα αλλά γνωρίζουμε ότι εργάζεστε σε πάρα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να το κανονίσουμε. Ίσως θα ήταν πολύ καλό να βρούμε έναν τρόπο να παρουσιάσετε εδώ όλες τις έρευνες και τις μελέτες σας. Γιατί είναι πραγματικά θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν τα μάλλα. Θέλω να σας θέσω και ορισμένα ερωτήματα μετά της ελπίδος ότι θα έχουμε κάποια ευκαιρία στη Βουδαπέστη να συνεργαστούμε και για τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Κάποια ερωτήματα και μονάχα. Για τη βία κατά των γυναικών. Υπήρχε διάχυτη ιδέα ότι το παρατηρητήριο για τη βία κατά των γυναικών θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον δικό σας φορέα. Έχετε κάτι σχετικά με το θέμα αυτό ή όχι. Γιατί πιστεύω ότι το ισπανικό μοντέλο, η παρακολούθηση των περιπτώσεων βίας γίνεται μετά από δικαστική απόφαση. Ενώ άλλες στατιστικές που συλλέγονται δεν αφορούν μονάχα τις περιπτώσεις που έχει προκύψει μια δικαστική απόφαση. Τι πιστεύετε λοιπόν για το θέμα αυτό. Έχουμε αρκετά συγκρίσιμα στοιχεία ή ου. Και ποιο είναι το μέλλον του θέματος αυτού. Θα έχουμε απλώς περιστασιακά συλλογή στοιχείων ή θα υπάρξει μια μόνιμη παρακολούθηση. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το εξής. Είπατε ότι σχεδιάζετε να προχωρήσετε και σε εκπαίδευση των ενδιαφερομένων. Σας ε, ενδιαφέρει η συμμετοχή στο σχέδιο αυτό που έχει να κάνει με την ε, διεύρυνση. Γιατί είχαμε κάποιους επισκέπτες οι οποίοι έλαβαν μέρος στο εγχείρημα άνθρωποι προς ανθρώπους. People to people δηλαδή. Θα ήταν πολύ σημαντικό και αυτό το σημείο της ε, ατζέντα να περιλάβει τη συνεργασία με τα άτομα αυτά που έρχονται από υποψήφιες χώρες. Και τε, εν τέλει θα, θα σας ρωτήσω πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε επαφή με τον φορέα σας, μεταξύ του φορέα σας και της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εισήγησή σας. Βρήκατε τώρα τη σωστή ερώτηση. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Έχω μία ερωτησούλα όσον αφορά τις προτεραιότητες. Ωραία όλα αυτά για τους ε, δείκτες και για τα στατιστικά όμως. Όσον αφορά αυτούς που τις αποφάσεις, χρειάζεται να γίνει μια συγκριτική μελέτη των δικαίων στην Ευρώπη. Και αυτό που είπατε για την βία, είπατε ότι θα κάνετε μια μελέτη για τις ε, πρακτικέ πρακτικές όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών. Πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτά να τα μάθει όλη η Ευρώπη. Το τι, είπατε, δεν κατάλαβα. Για την προτεραιότητα του θέματος γυναίκες και οικονομία και την τρόικα των προεδριών. Είπατε θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας ε, στο ρυθμό απασχόλησης, συγκερασμό δύο επαγγελματικού γυναικών κλπ. Όμως τώρα έφτιαξε ένα πλάνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια πρόταση τέλο πάντων όσον αφορά τις γυναίκες και τα κέντρα λήψη αποφάσεων και τις επιχειρήσεις, να κάτσουμε να δούμε επομένω τι ισχύει. Σε Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία. Τι θα κάνουν στην Ολλανδία. Να κάτσετε λοιπόν και να δείτε τι ισχύει όσον αφορά τη γυναίκα για τη λήψη των αποφάσεων και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και τι νομοθεσίε για να κάτσουμε να συγκρίνουμε. Εντύπωσή μου είναι. Όλες οι χώρες έχουν υπηρεστεί από την νορβηγική νομοθεσία. Υπάρχει επικάλυψη το θέμα γυναίκες και οικονομία, γυναίκες και λήψη αποφάσεων, γιατί βλέπετε ότι δεν ξέρει το ένα κράτος τι πει το άλλο. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Για τις άρεστες πρακτικές. Ευχαριστώ κυρία Τόμσον. Κυρία Μπαστός. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ισότητα των Φύλων. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι το έργο το οποίο φέρει σε πέρα αυτός ο φορέας και ποια είναι τα σχέδιά σας για τον επόμενο χρόνο σε σχέση με το έργο σας, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα αν προβλέπετε να υπάρχει συλλογή συγκρισίμων στοιχείων για το επιχειρήν μεταξύ των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα διάφορα κράτη-μέλη, εάν προβλέπετε κάτι τέτοιο, πότε θα έχετε τα στοιχεία αυτά για το επιχειρήν. Επίσης, σε σχέση με το συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αν γίνεται με εκτατικό τρόπο αυτή η συλλογή στοιχείων σε όλα τα κράτη-μέλη, και αν οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγών απόψεων μέσω του Ινστιτούτου αν έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την παρουσίασή τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κώστα. Ευχαριστώ κι εγώ. την κυρία ε, Είναι πολύ Είναι πολύ σύνθετη η δουλειά της, ε, γιατί και η αποστολή της είναι ιδιαίτερα χανής. Ε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για τη μέθοδο. Εσείς λέτε χρησιμοποιούμε αυτόν τον χρόνο για να βρούμε την μέθοδο εργασίας. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα και πρέπει να έχουμε φυσικά μια κοινή οπτική, διότι άμα, χάσετε, άμα έχουμε διαφορά στη μέθοδο τότε αλλάζουν όλα. Για τις στατιστικές, σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρώπης χρειαζόμαστε πιο εκλεπτισμένα, πιο επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία και εσείς είπατε ότι θέλετε να συνεργαστείτε σε δύο επίπεδα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα Ινστιτούτα τα οποία κάνουν ήδη αυτή τη δουλειά και σε εθνικό επίπεδο με τα εθνικά ερευνητικά συστήματα για να αποφύγετε και επικαλύψεις. Το gender mainstreaming πρέπει να περνάει μέσα από την Eurostat και εσείς θα πρέπει απλώς να κάνετε μετά πιο ε, μελέτες ε, πιο σε βάθος ε, με διάφορες θεματικές. Ουσιαστικά χρειάζεται το mainstreaming να βρίσκεται μέσα στην Eurostat. Δεν χρειάζεται εσείς να φτιάξετε μία στατιστική ε, βάση, διότι δεν έχετε καν τα κονδύλια. Πρέπει να εμβαθύνετε σε θεματικές που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Αλλά να ρωτιέμαι, αν εσείς συνεργάζεστε με τα ε, κράτη και δημιουργήσετε μόνιμα μόνιμα σημεία διαλόγου με τα διάφορα ε, τραπέζια διαλόγου θηλυκού γένους με τα κράτη-μέλη για να μπορέσετε να διαμορφώσετε τις στατιστικές σας. Πολλές φορές επίσης δεν έχουμε τα στοιχεία, το στοιχείο της ομοιογένειας. Μιλάμε εμείς ε, για εργασία και απασχόληση, λέμε αλλού 20%, 70% και δεν ξέρουμε αν είναι πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση. Το 2011 έχουμε δύο προτεραιότητες, οικονομία και περιβάλλον. Και εσείς λέτε όμως ότι για αυτά τα θέματα δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Τι εννοείται, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε, δεν υπάρχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες. Πώς επιλέγετε εσείς τους εμπειρογνώμονές σας όταν τους χρειάζεστε για να επεξεργαστείτε όλα αυτά τα στοιχεία. Τι αναφορές έχετε, πανεπιστήμια, μελέτες, για να δούμε και εμείς τη χώρα μας ποιοι είναι οι συνομιλητές μας. Και για τα μίντια, μη ε, ελληνιστή. πρόκειται για κάτι το δραματικό, το πώς δηλαδή μέσα από τα ΜΜΕ και δεν μιλάω μόνο για τη χώρα μου, την Ιταλία δηλαδή, περνάει η εικόνα της γυναίκας. Δεν μπορείτε εσείς να φανταστείτε να φανταστείτε να μαζέψετε και οπτικακουστικά ντοκουμέντα για αυτά τα φρικτά πράγματα τα οποία συμβαίνουν εις βάρος των γυναικών για να γίνεται και μια παρακολούθηση, ένα monitoring και να αναλυθούν και πρωτοβουλίες. Δεν μπορούμε εμείς να ασκούμε πολιτικές και μετά να διαψευδόμεθα από αυτό το οποίο γίνεται είτε συμβολικά είτε πολιτιστικά εις βάρος των γυναικών. Ευχαριστώ κυρία Κώστα. Έχω πολλούς, πολλές εγγεγραμμένες και θα ήθελα να τελειώνουμε μέχρι τις 6. Παρακαλώ να είστε σύντομες και να συγκεντρωθείτε στις προβληματικές μας για να υπάρξει και χρόνος, δηλαδή να απαντήσει η κυρία Λάνμπακ, η κυρία Νικόλα. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να χαιρετήσω αυτήν την συζήτηση σήμερα. Δεν έχω πολλές ερωτήσεις. γιατί είναι δύσκολο να καλυφθεί το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αυτού του κέντρου και δεν έχει νόημα να σας ρωτήσω για πάρα πολλές μελέτες. Και είσαστε ακόμα καινούργια σε αυτή τη θέση. Μία σύσταση απλώς θέλω να σας κάνω για μεγαλύτερη ορατότητα και αποδοτικότητα του Ινστιτούτου είναι καλύτερο να υπάρχει και ένας μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής μας και του δικού σας Ινστιτούτου. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαστε η επιστημονική, να αποτελείτε τη βάση επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης για την Επιτροπή μας και ίσως μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό για να σας πληροφορούμε για τα κύρια θέματα τα οποία μας απασχολούν και εσείς να μας δίνετε την επιστημονική πληροφόρηση για τα θέματα αυτά. Μια δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τη δραστηριότητά σας σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ημών. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι ότι η πολιτική για την ισότητα των φύλων δεν είναι πια πολιτική προτεραιότητα στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν μειώσει τις, ε, την υποστήριξη προς τα θέματα που ασχολούνται τα θέματα αυτά. Κλείνουν το Υπουργείο για τα γυναικεία θέματα, το κρατούν σε επίπεδο υφυπουργού μονάχα. Υπάρχουν κράτη-μέλη που ουσιαστικά ακυρώνουν τη, τη δυναμικότητα αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί στο μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε για να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μωρή Σαρτιέ, σας ευχαριστώ. Να επανέλθω κι εγώ σε ένα με ε, πρόβλημα μεθόδου. Είναι πολύ σημαντικές οι αναλύσεις σας για να τροφοδοτήσουν τις εργασίες μας. Λέτε ότι θέλετε να κάνετε στατιστικές που θα μας επιτρέψουν συγκρίσεις μεταξύ των κρατών. Θα ήθελα όμως να έχουμε και μία δυναμική ενόραση των πραγμάτων. Διότι πολλές φορές εμείς μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι προχωρούμε θετικά, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πολύ, κάνουμε, οπισθοχωρούμε πολύ σε σχέση με το, με, το παρελθόν. Θα ήθελα ε, για αυτό το θέμα της πρόοδου ή της οπισθοχώρησης, ε, της πισοδρόμησης, να μπορούμε να έχουμε στατιστικές για να παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρο. το το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, χωρίς μικρόφωνο κυρία Φιγκερέντου. Δεν δουλεύει αυτό το μαραφέτη. Χωρίς μικρόφωνο και πάλι κυρία Φιγκερέντου. Α, sí, Συγγνώμη. Απλώς θέλω να θέσω ένα ερώτημα που συνάπτεται με το θέμα της ε, διαφοράς της αμοιβέ ανδρών και γυναικών και με ορισμένε πρακτικές θετικού χαρακτήρα που έχουν ακολουθηθεί για να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Παραδείγματος το πρόγραμμα Equal όταν υπήρχε ακόμα οι σύμβουλοι ισότητος που υπάρχουν σε διάφορες επιχειρήσεις και επίσης αναφέρομαι σε ορισμένε μελέτες που έγιναν σε επιχειρήσεις όπου είχε εφαρμοστεί η πρωτοβουλία Equal για τη μείωση των ε, διαφορών αμοιβών στις επιχειρήσεις με το να μειώνεται ο αριθμός των βαθμών και κλιμακίων. Υπήρξε μια πολύ θετική λοιπόν εμπειρία στην Πορτογαλία για τα θέματα αυτά με συμμετοχή συνδικάτων, εργαζομένων και εργοδοτών, με αποτελέσματα τα οποία υπήρξαν αρκετά σημαντικά και θετικά σε μεγάλες επιχειρήσεις και οδήγησε αυτό επιχειρήσεις βιομηχανικού χαρακτήρα να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των γυναικών που εργάζονται στον τομέα αυτό, παραδείγματος χάρη στην αυτοκινητοβιομηχανία και να μειώσουν την ε, ψαλίδα σε επίπεδο αμοιβών που οδηγούσαν σε διάκριση κατά των γυναικών. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και μια καταγραφή τέτοιου είδους εγχειρημάτων στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να παρέμβουμε με πιο ενεργό τρόπο μέσω δράσεων οι οποίες θα οδηγήσουν στο να ξεπεραστεί αυτό το σκάνδαλο του να έχουμε αφενός μια οδηγία για την ισότητα αμοιβών, ενώ συγχρόνως παραμένει μια μέση διαφορά αμοιβών της τάξη του 18% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς προτίθεσαι να κάνεις στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Λάγκ Μπακ για να απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα. Σα ευχαριστώ για όλα τα ερωτήματα, τι ε, συστάσεις και τι προτάσει. Θα προσπαθήσω στη συντομία να απαντήσω πρώτα απ' όλα. Τα θέματα για τις μελέτες μας. Όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει πέρσι θα καταγράφονται πλήρως στην ετήσια μας έκθεση. Προετοιμάζουμε τώρα την ετήσιμη έκθεσή μας και θα υπάρχουν οι 67 συν 14 μελέτες, ίσον 81 με όλα τα ονόματα. Είναι πολύ χρήσιμο για σας να δείτε εσείς πώς έχουμε κάνει αυτές τις ε, μελέτες με στόχο την πρώτη συλλογή δεδομένων. Για το παρατηρητήριο. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε την αρχική σύλληψη του παρατηρητηρίου η απόφαση πρέπει να ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ύπαρξη στοιχείων συγκρισίμων. Ξέρετε ότι οι Ισπανοί έχουν συλλέξει μια σειρά στοιχείων για τη βία, αλλά προσπαθούμε και εμείς να δούμε με διάφορους τρόπους τη συλλογή αυτών στοιχείων για να μπορούμε να έχουμε κοινέ μεθόδους και συγκρίσιμα στοιχεία. Η πρώτη μας μελέτη θα είναι απλώς η απαρχή. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια μεγάλη ε, μελέτη. Είναι η υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα κάνει τη μεγάλη έρευνα στον τομέα αυτό. Συνεργαζόμαστε μαζί τους και θα χρησιμοποιήσουμε τα δικά τους δεδομένα για να ξεκινήσουμε να δούμε τι χάσματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά η πρώτη μας μελέτη είναι περιορισμένης εμβέλειας. Και μας ενδιαφέρει επίσης και η μελέτη για την για τις φέτες πρακτικές, ιδίως στην κατάρτιση, να δούμε πού μπορεί να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες για τα θέματα διεύνησης. Δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά η Γενική Διεύθυνση Διεύνησης μας προσήγγισε και φυσικά στον τομέα αυτό έχουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο στην εκπαίδευση. Θα έχουμε μία βάση δεδομένων και τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τα θέματα κατάρτισης για την ισότητα νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ και τη Γενική Διεύθυνση Διεύθυνσης. Και υπήρξαν και πολλά ερωτήματα για την ε, συνεργασία μεταξύ μας. Θα έρθετε να μας επισκεφθείτε το Μάιο, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Περιμένουμε αδειμόνως την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και να αναπτύξουμε και περισσότερη συνεργασία. Για τη διαφορετικότητα των νομοθετικών πλαισίων η μελέτη της οικονομίας, οι γυναίκες σε θέσεις ε, λήψης αποφάσεων, οι βέλτιστες πρακτικές όπως έλεγε η κυρία Τόμψεν για τις διαφορετικές ε, νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Αλλά το θέμα της οικονομίας και των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον όλες οι βέλτιστες πρακτικές θα βρίσκονται στη μελέτη αυτή την οποία θα ξεκινήσουμε το 2013 και αυτό θα το συζητήσουμε επίση όταν έρθουμε σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο γιατί εμεί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ συναρπαστική τρόποι αυτή, καθώ και προσέγγιση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και θα είναι επίση και μια πολύ καλή πρόταση τουλάχιστον για τι βέλτιστε πρακτικέ. να λάβουμε αυτό το θέμα υπόψη. Για τι γυναίκε επιχειρηματίε και τι βέλτιστε αυτών πρακτικέ. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τη συνεργασία με την Κομισιόν Γενική Διεύθυνση Επιχειρήν. Υπάρχει μια συνάδελφός μου η οποία είναι παρούσα σε ένα σεμινάριο για τα θέματα αυτά και θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς θα γίνει. Και η Γενική Διεύθυνση του Επιχειρήν θα συλλέξει και στοιχεία για τα θέματα αυτά και μεγάλη χαρά θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Στατιστικές και Ευρωστάτ. Έχουμε πολύ καλή στατιστική με τη Eurostat. Είναι παρόντες και στις ομάδες εργασίας μας. Ό,τι μελέτες και να κάνουμε, τις συζητάμε και με τη Eurostat, θα ήταν απώλεια χρόνου να μην χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά. Έχουμε και μια συμφωνία συνεργασίας μαζί τους. Για τους ερευνητικούς εν τέλει φορείς. Πώς τους επιλέγουμε. Ναι, αύριο μιλάμε τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα και θα συζητήσουμε για τη συνεργασία, τι μπορούμε να κάνουμε και μερικά από τα πράγματα τα οποία κάνουμε, τα οποία και αυτά μπορούν να είναι αντικείμενο συνεργασίας. Και υπήρχε και ένα ερώτημα για τους εμπειρογνώμονες, πώς τους επιλέγουμε. Ακολουθούμε την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ό,τι είναι αυτά τα οποία αναθέτουμε σε εμπειρογνώμονες θα πρέπει να γίνονται βάσει των κανόνων δημοσίων διαγωνισμών και έχουμε βέβαια προδιαγραφές, έχουμε συμβάσεις με πανεπιστήμια, είναι όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την αγορά εμπειρογνωμών. Για τα στερεότυπα ναι, θα παραμείνουν και θα δούμε τώρα πώς θα τα συμπεριλάβουμε στις μελέτες μας. Τα κράτη-μέλη και όσον αφορά το τι γίνεται με την ισότητα των φύλων και τις σχετικές περικοπές της πολιτικής. Αυτή δυστυχώ βλέπετε είναι η τάση που διαμορφώνεται, αλλά είναι κάτι που έχει εκφύγει των χειρών μα. Ε, βέβαια, θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε κάποιες προτάσεις, αλλά τελικά τα κράτη-μέλη possible... εξελίξεις, να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να διακρίνει κανείς κατά πού πάει το πράγμα, τι στατιστικά υπάρχουν και πραγματικά ε, τώρα έγινε το πρώτο βήμα. Γίνανε οι αρχικές μελέτες και επομένως αυτό το οποίο κάνουμε είναι μαζεύουμε από παντού. Δεν θέλουμε να, να στέλνουμε υπερβολικά πολλά στοιχεία μη στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι δύο-τρεις οι μελέτες σας γίνονται το χρόνο και έτσι θα μπορούμε να διακρίνουμε τάση και εξελίξεις. Τώρα, το μισθολογικό χάσμα και αρίστες πρακτικές. Φυσικά και εδώ πέρα είναι θέμα της Γενικής Διεύθυνσης για την απασχόληση. Ναι, ναι, ναι, έτσι μπορούμε να διακρίνουμε ποιες είναι οι καλύτερε πρακτικέ, οι άριστε πρακτικέ και επομένω να δούμε και τι γίνεται με τις ε, δημοσίευσει και επομένω προσπαθούμε να στηρίξουμε ό,τι γίνεται, ό,τι πρωτοβουλίες, ό,τι δράσεις γίνονται. Αλλά όλα αυτά για το μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Λάνμπακ. Εμείς ως Επιτροπή κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δημιουργηθεί αυτό το Ινστιτούτο. Είμαστε στο πλευρό σας. Και, περιμένουμε. και αναμένουμε βέβαια να έρθουμε και εμείς τώρα επίσκεψη στο Βίλνιους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 10. Η επιχειρηματικότητα των γυναικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ακούσουμε την εισηγήτρια την κυρία Γιανακουδάκη και έχετε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ να σας πω από πού ερχόμαστε και πού πάμε με αυτή την έκθεση. Μετά από πολλή έρευνα και είδα όλους αυτούς οι οποίοι πρόκειται από εταιρείε, ομίλους, ε, συνομοσπονδίες, συνεργάστηκα με την Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν, και τους ευχαριστώ και επίσης συνάντησα και τους σκιώδες, μου δώσαν και αυτοί ένα σωρό τι θέλει ο κόσμος, οπότε θα πρέπει να συνδούμε και άλλο με τους σκιώδες από πλευράς πάντως του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ε, θα πρέπει να έρχεται ο κόσμος να μου λένε τι γίνεται στα διαφορα κρατημέλη γιατί και εκεί υπάρχουν άριστες πρακτικές, όλα αυτά να τα βάλουμε στο κείμενο. Για να δούμε τώρα, ελπίζω όλα να βγουν στην παρουσίαση. Πρώτη διαφάνεια. Όχι, δεν προκύπτει. Όπου, α, μπορείτε να μπορείτε τώρα στο πρώτο slide δείχνει τι γίνεται με τους διάφορους συντελεστές τη απασχόλησης. Όταν μιλάμε για επιχειρηματίε, έχουμε ε, διαφορετικέ εκδοχές ε, ε, επιχειρηματικότητας. Είναι αυτοί οι οποίοι εκφύσεως είναι, λέει, επιχειρηματίες. Βέβαια αυτά τα μπαλάκια αυτοί που ό,τι και να γίνει θα καταλήξουν. Οι επιχειρηματίε είναι, είναι παίκτε ομάδα ή όχι. Με ενθουσιασμό, επομένω βουτάνε στα βαθιά. Και είναι και που δεν θα γίνουν ποτέ. Είναι αυτοί που θέλουν να δουλεύουν σε ένα δομημένο, διαδομένο περιβάλλον, αυτοί που σώφουν επομένω για επιχειρηματίες θα πρέπει να δούμε ποιοι μπορούν, ποιοι θέλουν να είναι. Και επομένω το σημείο κλειδί εδώ είναι αυτό που λέμε στην αρχή, ότι ε, εδώ δεν είναι θέμα φίλου. δεν μπορεί να είναι επιχειρηματία. Ούτε είναι θέμα παιδεία που έχει λάβει ο καθένα. Μου το είπε κάποιο σκιώδη. Εδώ είναι μόνο για του πολύ μορφωμένου. Όχι, δεν μπορεί να είναι επιχειρηματία. Πολύ νέο, ακόμα είναι στο σχολείο και πουλάει ζαχαρωτά στου μαθητέ του και αυτοί που έχουν απίστευτα διπλώματα, διδακτορικό κλπ. Και μπορεί να υπάρχει από διαφορετικέ για ζώνε, όλα αυτά δεν τα ξεχνάμε και. Επίση, πολλέ φορέ πρόκειται και για άντρε ή και για γυναίκε. Άλλο το σημαντικό για αυτήν την πρωτοβουλία είναι ότι είτε είναι άντρε είτε είναι γυναίκε, θέλουμε με αυτό το κείμενο να βοηθήσουμε τι γυναίκε να γίνουν επιχειρηματίε. Διότι, για κοιτάξτε, το 2, το 2, διαφάνεια 2, που δεν φαίνεται, το δύο που δεν βλέπετε ε, λέει ότι έχουμε λιγότερους επιχειρηματίες γυναίκες παρά άντρες. Και αυτό που προσπαθώ να δω είναι από τη βάση προς την κορυφή να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να έχουν την κατάρτιση, τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση. Επομένως, πώς θα προκύσουμε εδώ με ό,τι χρειάζεται τι γυναίκε. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι θα πρέπει επίση να προαγάγουμε τι καλύτερε πρακτικέ, θα πρέπει να συμβουλεύουμε τα κρατεί μελη με το πώς θα προχωρήσουν, πώς θα βοηθήσουν τις γυναίκες. Αυτό επομένως θέλουμε να ζητηθεί στην Επιτροπή μας για να αρχίσει το θέμα να, να συζητείτε. Επίσης, μπορούν να διαμετρήσουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ευελιξία, θα αποκτήσουν ισορροπία στη ζωή τους. Δεν είναι εύκολα αυτά. Γιατί κανείς όταν είναι επιχειρηματίας, 24 ώρες 24 ώρο πρέπει να δουλεύει. Παρακάτω. Ε, λέμε εδώ πέρα ότι έχουμε πάρα πολύ λίγε γυναίκε που είναι σε επιχειρήσει και λέμε ότι γενικά οι εργαζόμενε ε, πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Κυρίω γιατί ο βασικό του ρόλο είναι άλλο. Ε, Επομένω, αυτό που χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία στον επαγγελματικό του βίο και αυτό και που χρειάζονται περισσότερα δεδομένα. Για μα χρειάζεται να έχουμε γενικά δεδομένα για το τι γυναικών είναι αυτό, την εθνική προέλευση ηλικιακή ζώνη και όλα τα λοιπά. Το επόμενο. Και εδώ είναι η ουσία της έκθεσης. Λέει εδώ πέρα, μπορούμε να το κάνουμε. μπορούμε να αποκτήσουμε ό,τι χρειάζεται, μπορούμε και επομένω θα δώσουν τη μάχη τους και οι γυναίκες όπως και οι άντρες τουλάχιστον έτσι λένε. Από εκεί που έρχομαι εγώ και εδώ ε, μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα σχολεία, πανεπιστήμια, ειδικά μαθήματα και επίσης ε, τα πρότυπα. Γιατί αν έχουμε κάποια γυναίκα που είναι πετυχημένη θα πρέπει να τη δείξουμε. Παρέχουμε προσμήμεις και σε άλλες γυναίκες οπότε να τι εμπνεύσει και αυτέ να γίνουν το ίδιο. Ε, επιτυχίε, α πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο προβάλλουμε τη Μάργαρη Θάτσερ ή τη Βικτόρια Μπέκαμ μεταξύ των δύο προτιμάω ελαφρώ τη Μάργερ Θάτσερ, αλλά επομένω αυτό όμω είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορεί να εμπνεύσει. Καλά, σα αρέσει δεν μπέκαμε. Μπέκαμ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν βαριέστε. Εμπνέει. Ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Παρακαλώ. Υποστήριξη ε, από την ομάδα την κοινωνική που προέρχονται, οι μέντορες, οι οικονομικές πληροφορίες, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και πρέσβυρες, πρέσβυρες. Ε, τέλος πάντων η δουλειά που κάνει το η Κομισιόν και στο τέλος το τελευταίο το οποίο εξετάζουμε είναι επιλογή. Μπορεί κανεί να γίνει νέο, μπορεί να γίνει λιγότερο νέο, όταν έχει παιδιά, όταν δεν έχει παιδιά, να γίνει επιχειρηματία. Ανάλογα με πότε του έρχεται του και αυτό είναι το υπέροχο για αυτό το ρόλο. Μπορεί κανεί να διαλέξει, να είναι ευέλικτο, το, το, το, χρονισμό. Επίση είναι θέμα τεχνολογία αλλά και επικοινωνία. Σα το είπα πάρα πολύ γρήγορα διότι αυτό το οποίο πιστεύω θα το διαβάσετε. Το θέμα είναι τώρα που τελείωσα να πείτε εσεί τι σκέφτεστε. Σας ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση τη συναδέλφου. Δυστυχώ δεν έχουμε όμω χρόνο. Έξι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, αλλά σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι, δύο λεπτά το maximum. Θέλω να μιλήσω εξ ονόματος της Mary Χάνιβαου, γιατί δεν μπορεί να είναι παρούσα η Mary σήμερα. Λυπάμαι που δεν θα... Λυπάμαι που δεν μπορώ να με παρουσία σήμερα να ακούσω την πρώτη παρουσίαση της κυρίας Γιανακουδάκης για τις γυναίκες και τις μικρομισές. Θέλω όμως να ξεκινήσω ευχαριστών, ευχαριστούσα τουλάχιστον την κυρία Γιανακουδάκη για την υποστήριξη αυτής της έκθεσης και επειδή είναι τόσο επικοινωνική και τόσο καλά συνεργάστηκε με τους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η έκθεση αντιμετωπίζει ένα θέμα σημαντικής σημασίας και ένα θέμα που μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς μέσα στην οικονομική κρίση η οποία έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρηματογυναίκες, γιατί πολλές από αυτές δεν μπορούν πλέον να έχουν επιχειρήσεις. Για να έχουμε ανάκαμψη πρέπει τα κάτι μέλη να επενδύσουν πόρους σε αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα. Είχα ήδη την ευκαιρία <clears throat> ως και ότι για τα θέματα αυτά να συζητήσω με την κυρία Γιανακουδάκη και να της προσθέσω, να της προ προσφέρω μάλλον την ε, υποστήριξή μου. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση μπορεί με μικρές προθέσεις προσθήκες να βελτιωθεί. Όπως λέει η κυρία Γιανακουδάκη, τα κορίτσια μέσα από ειδική εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς λειτουργεί μια επιχείρηση όταν είναι ακόμα στο σχολείο. Είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθούν οι κοπέλες να βλέπουν μια ε, απασχόληση σαν επιχειρηματίες στο μέλλον και όσο πιο πολλοί το γνωρίζουν τόσο πιο πιθανό είναι ότι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν μια τέτοια καριέρα. Είναι απαραίτητο επίσης να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον στις κοπέλες όσο είναι νέες για να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους. Πολλές νέες κοπέλες ήδη αποθαρρύνονται από το να ασχοληθούν με το επιχειρήν γιατί το επιχειρήν παρουσιάζεται σαν μια καθαρά ανδρική απασχόληση. Πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για τις κοπέλες ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητε για να επιτύχουν στον τομέα αυτό. Έχω στείλει ήδη στην κυρία Γιανακουράκη κάποιες προτάσεις για τροπολογίες και θα παρουσιάσω και άλλες και προσλέπω σε μια περαιτέρω <clears throat> συζήτηση μαζί της. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορνέλσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θα ήταν θαυμάσιο πιο πολλές γυναίκες να γίνουν επιχειρηματίες και με σωστέ συνθήκες σε μια εποχή κρίσης όπου έχουμε πολύ μεγάλη ανεργία είναι πολλοί άνδρες αλλά και πολλές γυναίκες αυτοαπασχολούμενοι που προσπαθούν να βγουν έτσι από την κρίση και για τις γυναίκες είναι και μια λύση γιατί πολλές φορές η αυτοαπασχόληση σας δίνει την ευκαιρία να επιλέξετε καλύτερα τις ώρες εργασίας σας. Η έκθεση αναφέρει πολλά θέματα τα οποία είναι σημαντικά για να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την απασχόληση των γυναικών σε θέσεις επιχειρηματικές, καλύτερη γνώση, καλύτερη διαδικασία συμβούλευσης, πρόσβαση σε επενδυτικούς πόρους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο λείπει είναι η πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα, δικαιώματα σύνταξης, ε, ασφάλεια λόγω ε, αναπηρίας, ε, γονική <clears throat> προστασία και μέρημνα των παιδιών, γιατί σε πάρα πολλού χώρου. από πάρα πολλέ χώρε, μάλλον, η παιδική μέρημνα οργανώνεται από του εργοδότε, αλλά αν είναι κανεί αυτό απασχολούμενο, είναι πολύ δύσκολο να το εξασφαλίσει κανεί αυτό και είναι κάτι, ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να προσθέσουμε. Η έμφαση είναι για τα θετικά στην έκθεση της κυρίας Γιανακουδάκη, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και τα αρνητικά στοιχεία της ε, αυτοαπασχόλησης, όταν πολλές φορές οι γυναίκες υποχρεώνται να αυτοαπασχολούνται χωρίς να, τους, να το επιλέγουν, γιατί μια εταιρεία δεν θέλει να τους ε, καταβάλει κοινωνικές παροχές. Πρέπει επίσης να δώσουμε και μια προσοχή στις γυναίκες για τις οποίες η αυτοαπασχόληση θα μπορούσε να είναι μια λύση που εργάζονται παραγωγός χάρη στον οικιακό τομέα και ίσως θα είναι ενδιαφέρον να προσθέσουμε και κάτι για το πώς λειτουργούν τα τωρινά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν σε στόχο να τονώσουν το επιχειρήν, να κάνουμε μια έκθεση αντικτύπου για αυτά τα προγράμματα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και αυτό θα υποχρέωνε και ορισμένου οι οποίοι εργάζονται για τα προγράμματα αυτά να σκεφτούν και τη διάσταση του φίλου. Και για να κλείσω, κυρία Κιανακουδάκη, θα σας ευχαριστήσει ίσως ότι θα πάω τώρα στην ε, εναρκτήρια τελετή της, ε, του συνδέσμου των ε, δανών γυναικών, των ε, Ολλανδών μάλλον, γυναικών επιχειρηματιών, όπου θα επιλεγεί ένα νέο μοντέλο ρόλου για τον επόμενο χρόνο. Κύριε Μπάστους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μένω στον τον πιο σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιανακουδάκη για την προσέγγιση που επέλεξε. Και θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτά που είπε, να εστιαστούμε στα άτομα τα οποία έχουν τη δυνατότητα του επιχειρήν, είναι άνδρες και γυναίκες και ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Και πιστεύω ότι με την πρωτοβουλία αυτής της έκθεσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερες γυναίκες στο επιχειρήν. Αυτή είναι νομίζω η φιλοσοφία της εισηγήτριας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν οδηγεί σε μια καρικατούρα, σε μια γελιογραφία, ούτε στο να στιγματίσουμε τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο στο επιχειρήν. Απλώς πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκε στα κατημέλη, ώστε όλο και περισσότερες γυναίκες να είναι επιχειρηματίες. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση αυτή, η ανάγκη να υπάρξει περισσότερη πρόσβαση στην κατάρτιση και η δυνατότητα δημιουργίας δικτύων και η πρόσβαση στα δίκτυα πληροφορίας και επικοινωνίας, όλα αυτά παρουσιάζονται με τρόπο ο οποίο είναι πάρα πολύ σαφής. Αυτό όμως το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε πώς θα δώσουμε τις δυνατότητες σε όλο περισσότερες γυναίκες να γίνονται επιχειρηματίες. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι το σημείο της χρηματοδότησης είναι κομβικό και αυτό το αναφέρει πολύ σωστά η κυρία Γερακουδάκη. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι η εκπαίδευση για το επιχειρήν. Αυτή η εκπαίδευση για το επιχειρήν θα πρέπει να γίνεται ήδη στο γυμνάσιο και στο λύκειο και μετά φυσικά και στο πανεπιστημιακό επίπεδο και θα πρέπει να έχει ένα εγκάσιο χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια γενική μέρημνα για την εκπαίδευση των γυναικών προς το επιχειρήν. Τέλος, η δημιουργία επαγγελματικών δικτύων που ευνοούν την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και που δίνουν σε όλα τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πλατφόρμες που θα αρρωγούν τις γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν στον τομέα του επιχειρήν θα πρέπει να ενισχυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε και στον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας όπου χρειάζεται όπως ελέγχθη προηγουμένως από την πρόεδρο, από την διευθύντρια του Ινστιτούτου ότι χρειάζεται να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σέσκοβα. This is mine? Já Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα ήθελα να σας πω το εξή. Ίσως είμαι αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρηματίου, γυναίκας, μιας μη, μη ε, διότι πριν γίνω ευρωβουλευτήνα, όλη μου η επαγγελματική διαδρομή ήταν σαν επιχειρηματίας. Ήμουν σαν επιχειρηματίας, είχα μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ξέρω από μένους ότι πρόκειται πάρα πολύ καλά. να σας πω την απόψή μου. Σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξηγηθεί ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες πρώτον δεν χρειάζονται ιδιαίτερα κίνητρα ούτε πλεονεκτήματα. Αυτό το οποίο χρειάζονται είναι άλλο. Χρειάζονται σε επιχειρηματικό περιβάλλον και την αντίστοιχη νοοτροπία στην κοινωνία που ζουν. Ούτω ώστε να μπορούν να τα καταφέρουν, να μπορούν να συγκεράσουν οικογένεια και δουλειά. Και να μην κρέμονται από τον σύντροφο, σύζυγο κλπ. Já si myslím, že důležité je, abychom να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό και σας λέω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί αυτό στα κράτη-μέλη. Και όλα αυτά σας τα λέω από ιδία εμπειρία. Μάλιστα η κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Γιανακουδάκη. Δούλεψε σκληρά και είχε την καλοσύνη να λάβει υπόψη και τη δική μου άποψη. Βεβαίω. Και τα πράγματα τα λέει από βρετανική σκοπιά, όπω και εγώ. Ο φορέα των ΜΜΕ πρόβαλε ένα μανιφέστο στις τελευταίες εκλογές του 9 Έκλεισε προς εμάς, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και έλεγε σταματήστε την πολυνομία. Όχι άλλους νόμους. Άρα, τι να την κάνουν αυτή την οδηγία. Γιατί υποφέρουν οι ΜΜΕ. Είναι πιο μεγάλη εργοδότες στη χώρα. Υπάρχει πολυνομία, η υπερβολική, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό επαναλαμβάνω συνέχεια. Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Είδαμε τη ΠΕΤΟΔΕΚ για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Έχω πάρει ένα σωρό επιστολές από ψηφοφόρους μου και λένε μην ξεχνάτε ότι τα ασφάλιστα δεν θα μειωθούν. Μα όχι των, γυναικών Η, ομιλήτρια. Θα ανεβάσουν των γυναικών στο επίπεδο των ανδρών τα ασφάλιστρα. Άρα, πού να ωφεληθούν Δηλαδή όταν υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι τελικά αυτό ε, είναι χαστούκι στι γυναίκε. Δεν επηρεάζει του άντρε. Επομένω, όλα αυτά για μένα είναι απαρχαιωμένα. Πάνω να βρείτε καινούργιο πρότυπο και ξαναγείτε στο μοντέλο τη δεκαετία του 70. Δείτε λίγο πιο ψύχρεμα, πιο νυφάλια. Αυτό που χρειάζεται είναι να φτιάξετε θέσει εργασία για όλου. Άρα παρακαλώ σταματήστε να θεσπίζετε νέα νομοθεσία. Ευχαριστώ κύριε Νικολάη. Ευχαριστώ πρόεδρε που έχει περάσει ώρα και για αυτό έχω να σας πω ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε τώρα ολόκληρη συζήτηση για την έκθεση, αλλά απλώ θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την συγκίτρια και από αυτήν την έκθεση θέλουμε να απαντήσει εις δύο ερωτήσεις. Ο κάτω άντρα για μια δουλειά είναι η γυναίκα. Ισχύει ή όχι. Επίσης, κάτι πρέπει να γίνει όσον αφορά τις ΜΜΕ. Θα πρέπει να προβάλλουμε κάποια πρόταση, κάποια μέτρα να μπουν στην επιχειρηματικότητα οι γυναίκες. Τώρα που σοβεί η κρίση και που έχουμε αυτή την τρικυμία στην αγορά απασχόλησης. Τέλος πάντων, έχουμε σκεφτεί κάποιες τροπολογίες και θα τις υποβάλουμε στην συγκήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Γιάννα Κουδάκη που έχει εκφράσει τις ιδέες της με μεγάλη σαφήνεια και εξάλλου με την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα <clears throat> μεταξύ μας. Γιατί πριν από τρία χρόνια είχαμε κάνει μια έκθεση για τη συμμετοχή των γυναικών στη βιομηχανία που είχα σταθεί εγώ εισηγήτρια. Και είχε μεγάλη σημασία τότε αυτή η έκθεση στο παρελθόν για να καταδείξει τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον τομέα της βιομηχανίας, τις τεράστιες διακρίσεις που υπάρχουν μεταξύ και γυναικών και η έλλειψη πρόσβαση σε ορισμένες σε ορισμένους κλάδους βιομηχανικούς που θεωρούνται <clears throat> ανδρικοί και γι' αυτό αναφέρθηκα και στο πρόγραμμα Equal <coughs> προηγουμένως και επίσης υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα σε μια δύσκολη εποχή όπως αυτή να δώσουμε προσοχή στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν επικεφαλής τους γυναίκες. Αν έχουν προβλήματα αυτές οι επιχειρήσεις σήμερα, έχουν πολύ μεγαλύτερες ε, δυσκολίες όταν ε, βρίσκονται επικεφαλής τους γυναίκες, γιατί έχουν μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση που αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερο δισταγμό τις ε, γυναίκες οι οποίες διαχειρίζουν αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε έμφαση στο σημείο αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω και πάλι να συγχαρώ λοιπόν την ε, κυρία Γιάννα Κουδάκη παρά τις δυσκολίες που έχουμε, τις διαφορές που μπορεί να έχουμε σε ιδεολογικό πλαίσιο υπάρχουν στοιχεία εδώ τα οποία θέλω να υποστηρίξω και άλλα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να βελτιώσουμε, ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ, και η Πρόεδρος. Η Αντιπρόεδρος, η κυρία Μογά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και στο ύφος και στη μορφή και στην ουσία. Δεύτερο, πρέπει να επιμείνουμε στην ανάγκη του να συνοδεύουμε τα δίκτυα γυναικών με πολιτικές εγκύτητας. Οι γυναίκες επιχειρηματίες χρειάζονται να υποστηρίζονται μεταξύ τους, όχι μόνο με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο να δημιουργούνται δίκτυα γυναικών ή επιχειρηματιών τις οποίες μπορούμε και εμείς να υποστηρίζουμε με μεθόδους παρενάζ αιγίδας. Επίσης, οι γυναίκες θα έπρεπε να αρχίσουν να συμμετέχουν περισσότερο στα τοπικά εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, τα οποία πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν γυναίκες διότι συνήθως τα βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια ψάχνουν κυρίως τους άντρες θεωρώντας ότι ξέρουν καλύτερα τα πράγματα από ότι οι γυναίκες. Πρέπει να αρχίσουν λοιπόν να ψάχνουν και γυναίκες. Τα τοπικά επιμελητήρια πρέπει να αρχίσουν να πηγαίνουν προς τις γυναίκες διότι οι γυναίκες ξέρουν πολύ καλύτερα τι κάνουν. Εκπρόσωπος της Κομισιόν έχει το λόγο. Thank you very much, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτή την έκθεση και ευχαριστεί πολύ την κυρία Γιάννα για τη συνεργασία. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Έχουμε μια δημοσίευση που κάναμε σήμερα για πρόσκληση ενδιαφέροντος σε σχέση με τις γυναίκες που ασχολούνται με το επιχειρήν. Αν θέλει κανείς λοιπόν ως εμπλεκόμενος να συμμετάσχει θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης για το πρόγραμμα των γυναικών πρέσβεων έχουμε 70 πρέσβης σε 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μοντέλα ρόλου για το επιχειρήν και έχουμε και τον έρασμο για τους νέους επιχειρηματίες 42% είναι γυναίκες και αυτό είναι πρόγραμμα ανταλλαγής επιχειρηματιών μεταξύ των χωρών μεταλαμπάδευσης 42% του προγράμματος γίνεται με τις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Και τώρα οι διερμηνείς θέλουν να πάνε σπίτια τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εργασία, λέει η πρόεδρος. Και η κυρία Γιάννα Κουδάκη μπορεί να κάνει τις τελευταίες παρατηρήσεις και μετά συνεχίζουμε στην σεξπυρική γλώσσα χωρίς διερμηνία. Κυρία Γιανακουδάκη, έχετε τον λόγο. Και ευχαριστώ τους διερμηνείς. I'll be, I'll be very quick. Um, I'd like to thank all, all the kind comments actually um, and just say that this is a work in progress